Okay, colleagues, I think we're going to make a start. Συνάδελφοι, νομίζω να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Με συγχωρείτε που καθυστερήσατε λίγο. Αν είστε σαν και εμένα, θα Σα έκανε εντύπωση ότι έχουμε συνεδρία σε αυτήν την αίθουσα. Συνήθω είμαστε στο άλλο κτίριο και έπρεπε να περπατήσουμε και όλο αυτό το δρόμο. Τέλο πάντων, να ξεκινήσουμε αμέσω γιατί έχουμε καθυστερήσει και έχουμε και προσκεκλημένου και να περάσουμε στο πρώτο θέμα τη ουσία, επί τη ουσία ε, πολύ γρήγορα. Πρώτο σημείο λοιπόν, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Όπω ε, σα υποβλήθηκε, μπορούμε να την ε, εγκρίνουμε. Σημείο 2. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση στι 10 και 11 Ιουλίου η Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών οργανώνουν την ε, συνεδρίαση για την αποκεντρωμένη διαχείριση με 600 συμμετέχοντες από τις ε, τοπικές τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Χωροσακία και την Λατινική Αμερική. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι θέλουμε να ελοπίσουμε ε, την συμφωνία για τους στόχους τη χιλιετίας, για τη βιώσιμη ανάπτυξης και το πρόγραμμα μοιράζεται τώρα που μιλάμε. Όποιοι θέλουν να συμμετάσχουν είναι ευπρόσδεκτοι. Επίση, να σα ενημερώσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο έχουμε συνεδρίαση επιτροπής. Δεν προβλεπόταν ε, στο πρόγραμμα του έτους. Ε, προγραμματίστηκε για Δευτέρα το βράδυ στις 8 η συνεδρίαση. Ψηφοφορία για σημαντικά θέματα για το EFSD, ε, που ελπίζω να έχουμε επιτυχή διάλογο σήμερα και ενδεχομένω για την οικοδόμηση δυνατοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Αυτά τα δύο σημεία θα ε, ψηφιστούν. Θα λάβετε την ημερήσια διάταξη αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Και θα τα δούμε στο Στρασβούργο στις 8. Με συγχωρείτε, η συνεδρία τη Επιτροπή θα ξεκινάει 7.30, 8 θα είναι ψηφοφορίε. Δύο ξεχωριστέ λοιπόν συνεδριάσει. Ε, στην πρώτη φάση κοινή συνεδρίαση με τι εξωτερικέ υποθέσει, μετά με την Επιτροπή Προλογισμού ε, και μετά μόνοι μα. Δύο συνεδριάσει ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε στις 7.30. Θα ενημερωθείτε. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών 25 και 26 Ιανουαρίου, 24 και 25 Απριλίου και 3 Μαΐου. Εάν έχετε παρατηρήσεις, παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία στο τέλος της συνεδρίασης. Ιδάλλως θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Σημείο 4. Για την συνεδρίαση των συντονιστών 30 Μαΐου απόφαση. Και αν πάλι δεν υπάρξουν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν. 5 Επιτροπή, έχετε τίποτα να μας πείτε. Έχετε ανακοινώσει. Όχι, να θυμίσω στους συντονιστές ότι θα συναντηθούμε ε, για πρωινό στις 8. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε ποιος θα έρθει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να περάσουμε στο σημείο 6. Έκθεση για την αποστολή παρατηρητών στην Γκάμπια τον Απρίλιο. Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, είμαι βέβαιο ότι η Τζιν θα μας δώσει το ιστορικό, αλλά μιλάμε για 22 χρόνια πολιταρχικού καθεστώτος με τον πρόεδρο Γιαχαγιάμε, ο οποίος ε, τον Δεκέμβριο υπτήθηκε από τον Ανταμπάρο αλλά η Τζιν ξέρει πολύ περισσότερα, είτε καλύτερα να μας τα πει. Τζιν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Παρότι ήταν μόλι ε, στι αρχέ Απριλίου, φαίνεται να έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Ίσως επειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο ξέρετε ότι είχαμε και άλλε εκλογές και έτσι είχαμε άλλα στο μυαλό μας. Όμω ε, αυτέ οι εκλογέ ε, στην Γκάμπια έχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα. ο επικεφαλή ε, της ε, αποστολή μας ήταν ο Δεν έχουμε ακόμα τελική έκθεση από εκείνον. Έχουμε όμως μια σύντομη έκθεση από ε, την κυριοβουλευτική αποστολή παρατήρηση εκλογών. Είχαμε λοιπόν μια εξαμελή αποστολή από έξι χώρες και τέσσερι πολιτικές ομάδες. Η κυρία Κέγγε που είναι σήμερα μαζί μας. Πήγαμε λοιπόν για αυτέ τι τρει-τέσσερι ημέρε, μικρό το διάστημα για να παρακολουθήσουμε τις ε, εκλογές και τη διενέργειά τους. Συναντηθήκαμε με ε, διάφορα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, μία σειρά πολιτικών κομμάτων, πολιτικών ηγετών, δύο από των οποίων ήταν και υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και αυτό ήταν ε, μια Αυτές, εκείνες οι εκλογές ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσε, γιατί όπως είπε και η Πρόεδρος, τότε είχαμε αυτά τα 22 χρόνια, όλο και πιο αυταρχικής παρουσίας ε, του ε, Προέδρου για με, όμως ε, κάτι το οποίο θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι έκανε και τις εκλογές το Δεκέμβρη και τελικά είχαμε μια επτακομματική συμμαχία, ένα συνασπισμό που αντιτάχθηκε σε εκείνον και κέρδισε τις εκλογές. Ο νέος Πρόεδρος, ο κ. Μπάρου, που ε, και στο παρελθόν ήταν ε, στο Λονδίνο και τώρα βρίσκεται αυτοεξόριστος. Έχει κερδίσει λοιπόν ως υποψήφιος, έλαβε πάνω από το 43% ε, των ψήφων, ο πρόεδρος 39,6% και είχαμε και ένα τρίτο ψήφιο που πήρε περίπου το 17% των ψήφων των έγκαιρων σύμφων. Οπότε ήταν ε, μάλλον αναπάντεχο το αποτέλεσμα και μετά στις γενικές εκλογές είδαμε, στις βουλευτικές δηλαδή, πρώτο το, να δούμε κατά πόσο ε, ο συνοσπισμός, ο περσινός του 16 θα κρατούσε. Έχουμε ακόμα και πέντε μέλη του Κοινοβουλίου ε, που ε, ορίζονται από τον ε, Πρόεδρο ή αν δεν θα έστεκε τελικά αυτός ο συνασπισμός και τελικά θα έσπαγε. Σε περίπτωση που δεν κατέληγαν σε συμφωνία για μια γενική συνεργασία, είδαμε κάποιες μερικές συμφωνίες σε, μεταξύ των μελών αυτού του προηγούμενου συνασπισμού και θεωρούμε ότι αν υπήρχε περισσότερο χρόνο, περισσότερη βούληση, θα είχαν καταλήξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα με περισσότερε έδρε τελικά. Ε, τελικά όμω το UDP που θεωρείται το κόμμα του Προέδρου θεωρείται το μεγαλύτερο κόμμα. Και έτσι θεωρούσαν ότι ε, θα μπορούσαν να δεχθούν περισσότερες έδρες ε, υπό μια συμφωνία. Τελικά όμως υπήρχε ε, μια δικογνωμία σε πολλέ έδρε και επειδή είχαμε αριθμό ρεκόρ υποψηφίων, 239 υποψήφοι, μεταξύ των οποίων κάποιοι ανεξάρτητοι, στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες. Και το εκλογικό σύστημα της Γκάμπια είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν έχει τυπωμένα ψηφοδέλτια, Ουσιαστικά έχουμε ένα τύμπανο ανεποψήφιο στα χρώματα του πολιτικού κόμματος. Σε κάθε ένα από αυτά τα τύμπανα στο βάθος βλέπει κανείς, βρίσκει κανείς ένα ε, λίγη άμμο. Υπάρχει και μία καβάνα και τους δίνει κάποιος έναν ε, βόλο, πηγαίνει μέσα στο... Ε, να ψηφίσει τέλο πάντων ε, με τον βόλο αυτόν και το ρίχνει ε, στο αντίστοιχο τύμπανο με το όνομα του υποψηφίου. Ρίχνει κάποιος λοιπόν το βόλο μέσα στο τύμπανο. Ακούγεται η καμπάνα και έτσι ξέρουμε ότι έχει ψηφίσει κανείς. Ιδιαίτερα λοιπόν αυτό το σύστημα και ιδιαίτερα το παρουσιάζει και σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους. γιατί στο τέλος ε, βγάζουν την ε, ε, σφραγίδα ασφαλείας, αναποδογυρίζουν τα τύμπανα, βγαίνουν οι βόλοι, μπαίνουν σε ένα πλέγμα που παίρνει περίπου 200 βόλους. Όλοι το κοιτάζουν αυτό το πλέγμα και δηλαδή εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και το καταξύ των πολιτικών κομμάτων. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι 200 οι βόλοι, τους ξαναβάζουμε στο τύμπανο και βγαίνουν μετά οι υπόλοιποι. Είναι λοιπόν πολύ γρήγορη η μέθοδος καταμέτρησης, αρκεί να μην πέσουν κάτω οι βόλοι. Οπότε είναι γνωστοί οι αριθμοί Είναι πολύ διαφανές ε, το σύστημα, εξαιρετικά σαφές, ιδίως για μια χώρα που δεν έχει υψηλά επίπεδα αλφαβητισμού. Οπότε έχουμε την αίσθηση ότι εντάξει βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα, δεν μπορεί κάποιος να ψηφίσει ε, από το εξωτερικό και μάλιστα υπάρχει σημαντικό ε, ποσοστό Γαμπιανών που διαμένουν στο εξωτερικό, δεν μπορεί κάποιο να ψηφίσει εκ των προτέρων. Όπω και να έχει, είναι ένα πολύ σαφέ και διαφανέ σύστημα, εύληπτο και πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό. Σε αντίθεση με άλλες εκλογές ε, στις οποίες έχουμε συμμετάσχει ως παρατηρητές. Βέβαια, εντάξει, εδώ μετράει και το γεγονό ότι στη Γάμπη έχει πολύ μικρό πληθυσμό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον πληθυσμό ακριβώ. Ίσως 800 ψηφίσαντε σε ανεκλογικό κέντρο. Οπότε δεν είναι και τεράστιο αριθμό των ψηφοφόρων συνολικά. Εμείς ε, Λοιπόν, ήμασταν σε 40 εκλογικά κέντρα, τρεις ομάδες. Εγώ έμεινα στην Παντζούλη, στην ε, πρωτεύουσα. Άλλοι πήγαν αλλού, σε άλλε πόλει η ομάδα. Τώρα, για τα άλλα ζητήματα που παρατηρήσαμε εκεί, Είχαμε έναν αριθμό ρεκόρ υποψηφίων, αλλά όχι γυναικών υποψηφίων. 20 τον αριθμό ήταν οι γυναίκες και μόλις τρεις εκλέγησαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε θίξει ε, και στις επαφές μας με τα πολιτικά κόμματα και με τις οργανώσεις ε, που εργάζονται ακριβώ ε, για την ε, ανάπτυξη και την υποστήριξη της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, είπατε και εσείς, Πρόεδρε, ότι είναι αρκετά καταπιαστικό το καθεστώς. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ε, ιστορικά και παραδοσιακά είναι ισχυρά τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό όμω συμβαίνει σιγά-σιγά στη Σενεγάλη και σε άλλες χώρες τώρα θεωρούν ότι έχει νόημα να έχει κανείς έναν ε, αντιπρόσωπο στην ε, Γκάμπια, γιατί έχει νόημα να έχουν εικόνα από τα όσα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, ούτως ώστε ο κάθε υποψήφιος να έχει χρόνο ομιλίας για να παρουσιάσει τις θέσεις του αν και υπήρχαν δυσκολίες, ε, περιορισμένος χρόνος, ε, πολύ δύσκολες μετακινήσεις μέσα στη χώρα και πολύ περιορισμένος εξοπλισμός. Έκαναν λοιπόν σημαντικές προσπάθειες. Οι περισσότερες πληροφορίες ε, αυτές μεταδίδονται μέσω ραδιοφώνου και σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις πιάστικες περιοχές. Μέσα ενημέρωση λοιπόν είναι ένα από τα ε, στοιχεία στα οποία θα υπάρξει σημαντική εξέλιξη στο μέλλον. Τώρα, για τα αποτελέσματα, το UDP νίκησε με 31 εκλεγμένους υποψηφίους, τα κόμματα του συνασπισμού τα πήγαν και αυτά πολύ καλά, με ακόμα 11 θέσεις που πήγαν σε τρία κόμματα που ήταν ε, μέλη ε, του Σασουσμού του 16. Ε, το κόμμα του πρώην Προέδρου κέρδισε πέντε θέσεις στις παραδοσιακές εκλογικές περιφέρειες. Και το τρίτο κόμμα στις προεδρικές εκλογές, το 17%, είναι το μοναδικό κόμμα που ορίζει υποψηφίου σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και κέρδισε και αυτό πέντε τέτοιες ένδρες. Έχουμε λοιπόν ένα πολυμελές ε, και πολυπρόσωπο κοινοβούλιο, αλλά με ξεκάθαρο νικητή. Πρέπει να δούμε τι πόρους μπορούμε να διαθέσουμε για να συνεργαστούμε με αυτό το νέο κοινοβούλιο. Προκειμένου να λειτουργεί πραγματικά ως κοινοβούλιο, ε, να υπάρχει πραγματική ε, λογοδοσία και έλεγχος, Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πρόκληση από εδώ και πέρα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία θα θέλω να σταθώ. Αλλά έχουμε και συναδέλφους που συμμετείχαν και εκείνοι στην αποστολή. Και ευχαριστούμε πολύ και το επιτελείο μας που μας ακολούθησε, γιατί τελικά όλα πήγαν καλά και υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Thank you very much, Jean. Um, I don't Σας ευχαριστούμε. Jean. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να πει η Σεσίλ Κιέγγε για την αποστολή. Θέλει. Παρακαλώ, Σεσίλ. Ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώ την Τζιν Λάμπερτ για τη δουλειά που έκανε ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Διότι εργαστήκαμε εξαιρετικά μαζί. Τα σημεία που τώρα μας ε, ανέφερε με βρίσκουν σε όλα σύμφωνοι. Ήταν ε, δουλειά πολύ σημαντική και παρακολουθήσαμε την ιδιαιτερότητα του συστήματος που ψηφίζουν οι άνθρωποι εκεί και του συστήματος ε, μιας της μετάβασης από μια δικτατορία σε ελεύθερες εκλογές πρώτη φορά που να ελεύθερε εκλογέ στη χώρα. Ε, να προσθέσω απλώ μια παρατήρηση δική μου, δύο μάλλον παρατηρήσει, τη δική μου συμβολή. Η δυνατότητα που είχαν οι δικαστικέ λειτουργοί, γυναίκε δικαστικέ λειτουργοί και που ζητούσαν υποστήριξη στη δουλειά του είναι σημαντικό για να υπάρχει ανεξαρτησία κυρίω για το συνταγματικό δικαστήριο. Ε, το οποίο ε, και όταν μέχρι πρόσφατα από δικαστές άλλων χωρών. Πραγματικά μας ε, συγκίνησε η δύναμη χαρακτήρος και η τόλμη των ε, γυναικών αυτών. Και όπως είπε και η Τζιν, πρέπει να τη στηρίξουμε. Πρέπει να τη στηρίξουμε γιατί είδαμε γυναίκες να είναι δυνατές και να έχουν τη δυνατότητα και για να αντιδράσουν. Το άλλο που θέλω να πω είναι κάτι που δεν έχει ε, σχέση με την αποστολή μας επιτόπου, αλλά ενδιαφέρει την, αποστολή, την επιτροπή μας εν γέννη. Ακόμη και αν η Γκάμπια είναι μια μικρή χώρα στην Ήπειρο αυτή, έχουμε πάρα πολλούς ε, πρόσφυγες. Και στην ε, πορεία τους πρέπει να προσφέρουμε κάποια υποστήριξη, κάποια συνοδεία. Δηλαδή να φροντίσουμε και την ένταξή τους εδώ, αλλά και την ένταξή τους εκεί. Αλλά ενισχύοντας τη δική μας τη συνεργασία προς τη συγκεκριμένη χώρα. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Θα ήθελαν να ζουν σε μια χώρα που να λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Κάμπια να περάσει με επιτυχία από αυτή τη μεταβατική περίοδο. Γιατί βγαίνει τώρα από ένα πολιταρχικό καθεστώ, μια δικτατορία. Και είναι πολλοί πρόσφυγε για να έρχονται από μια τόσο μικρή χώρα, τόσο πολύ άριθμοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Χέιντι. Ευχαριστώ. για αυτήν την ε, πολύ ευχάριστη εκλογική διαδικασία και την πολύ ευχάριστη ενημέρωση. Ανέφερε, Τζιν, ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να στηρίξει την ε, οικοδόμηση δυνατοτήτων στη χώρα αυτή. Αυτή ήταν η τελική σου δήλωση και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και όλα τα σχετικά. Πώς Αξιολογείς εσύ τη δυνατότητα να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στο κράτος δικαίου σε όλες τις περιοχές. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ μια-δυο ερωτήσεις. Το τι θα γίνει μετά είναι ένα θέμα, διότι προφανώς εδώ αποφύγαμε μια καταστροφή, ε, οι εκλογές οργανώθηκαν, θα μπορούσε να είναι άλλο ένα αποτυχημένο κράτος, αλλά αποφεύθηκε σύγκρουση που δέχτηκαν οι σειράξει στη χώρα αυτή, το θέμα είναι πώς θα κάνουμε το σύστημα πιο ανθεκτικό. Τι έκανε όμως αυτή τη φορά να αντέξει το όλο σύστημα, η στήριξη της διεθνούς κοινότητας, πώς θα μπορέσει να έχει μια ειρηνική μετάβαση η χώρα αυτή σε ένα άλλο σύστημα και πώς γίνεται να είναι πάντα οι εκλογές έτσι φιλιρινικές. Και ω προ την πολιτική αντοχή και αντεκτικότητα, δεν μα ενδιαφέρει μόνο η πολυοικονομική οικονομική του αντοχή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η οικονομική ακριβώ ενθεκτικότητα, διότι η Γκάμπια είναι μια χώρα που τη γνωρίζουμε πολύ καλά από τη δικιά μα χώρα, γιατί είναι ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό για του δικού μα πολίτε. Εδώ λοιπόν είμαι βέβαιη ότι θα ενημερώθηκε για τον αντίκτυπο στην οικονομία από την πολιτική κρίση, παρόλο που η επίσκεψη ήταν πολύ σύντομη σε διάρκεια. Υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε για να. Εντάξει, είναι μικρή χώρα η Γκάμπια αλλά μπορούμε να φροντίσουμε να είναι ανθεκτικοί και στο μέλλον. Σε άλλες χώρες που έχουμε εξετάσει στην Επιτροπή μας, ε, μάλλον αυτή τη χώρα δεν έχουμε εξετάσει όλη φορά στην Επιτροπή μας, από το εγώ πρόεδρος τουλάχιστον. Ακούστε. Αυτό που είπε η Σεσίλ για το δικαστικό σώμα. Είναι σημαντικό πραγματικά η εντύπωση αυτή ότι το δικαστικό σώμα ενώ είναι ε, για την Κάμπια και προέρχονται δικαστές από την Κάμπια, δεν λειτουργεί, δεν αποδίδει δικαιοσύνη. Και συνεννοηθήκαμε, μάλλον συζητήσαμε ανθρώπου από το δικηγορικό ε, σύλλογο ε, και υπάρχουν εκεί μάλιστα γυναίκες πάρα πολύ δυναμικέ που θα τις στέλαμε πραγματικά υπήρχε ανοιχτό πνεύμα θέλουν να μας υποστηρίξουν. Within the country, because they recognize how... Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα, γιατί φαίνεται ότι το πρόβλημα αυτό γίνεται χρόνιο με τους λειτουργούς ε, της δικαιοσύνης ε, και σε ό,τι αφορά σημαντικές ανησυχίες που προκύπτουν. Άρα πράγματι είναι σημαντικό να στηριχθεί το δικαστικό σώμα. Μπορεί να γίνουν ε, να έγιναν ειρηνικά οι εκλογές. Βέβαια ένα κόμμα θα προσβάλλει από ό,τι είπε Υπήρξαν κάποια άλλα ζητήματα με την ε, προληπτική στρατεία του Προέδρου σε διάφορες περιοχές της χώρας κτλ. κτλ. Επισκέψεις τέλο πάντων του Προέδρου. Γιατί θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι κάνει καμπάνια με αυτές τις επισκέψεις ο Πρόεδρος. και θα είναι τα πράγματα ε, χειρότερα την επόμενη φορά, πιστεύω. Δηλαδή θα υπάρξουν και άλλοι που σας προσβάλλουν σε εκλογή. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί η δικαιοσύνη να αποφαίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει επίσης να υπάρχει εμπιστοσύνη στο εκλογικό σύστημα και στην ανάπτυξη των θεσμών στη χώρα. Αλλιώς γιατί να επενδύει κανείς αν θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και όλα γίνονται όπως τα θέλει ο Πρόεδρος. Μερικοί μας είπαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσει ο πρόεδρος η εταιρεία, για παράδειγμα, η ΤΑΔΕ, η ΔΙΝΑ δεν εκπλήρει κάποιους κανόνες, όπως έγινε πρόσφατα, μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο, σε δυσχερή θέση εν λόγω επιχείρηση. Um, Πράγματι λοιπόν για να υπάρχει και επενδυτική εμπιστοσύνη αυτό είναι σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την τουριστική, τον τουριστικό κλάδο. Εντάξει, καλά είδαμε να πάνε τα πράγματα, όμως το θέμα είναι να μην προκαλείται βλάβη στο περιβάλλον. Ορισμένοι που είναι στην αντιπολίτευση τώρα έχουν εκφράσει καταγγελίες και προβλήματα που υπάρχουν με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεν γίνονται οι απαιτούμενες προσπάθειες για την προστασία της χλωρίδας της πανίδας και την προστασία του περιβάλλοντος. Σίγουρα πρέπει να προστατεύσουν την τουριστική δραστηριότητα από την οποία πολύ και η γεωργία επίσης είναι ένα θέμα. Υπάρχουν καλλιέργειε στη χώρα, σημαντικές και είναι καλό να αναπτυχθεί η γεωργία και σε σχέση και με, την, με τον τουρισμό όπως είπα. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθούν οι απαραίτητε υποδομέ και αυτό μας το είπαν στην εκεί μα επίσκεψη. Με την αλλαγή Προέδρου ε, θα μπορούσε να προκύψει και κάποια άλλη αλλαγή, δηλαδή να νιώσει ο κόσμος ότι μπορεί να αναπνεύσει, ότι είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Και νομίζω στην ε, προσέλευση το 42% πήγαινε να ψηφίσει στις βουλευτικές, στις σε μεγαλύτερο το ποσοστό. Βέβαια πρέπει να αναπατριστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου, αλλά τέλος πάντων. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία και ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν, θα βελτιωθούν. Πρέπει λοιπόν να υποστηριχθούν οι μηχανισμοί και για την ενίσχυση του κράτους δικαίου των μέσων επικοινωνίας ε, των κοινοβουλευτικών θεσμών. Αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα για να υπάρξει πραγματικά διάρκεια στην ε, αλλαγή της διάθεσης και στην ε, εμφάνιση αυτή της αισιοδοξία που αλλιώ θα εξανεμιστεί σύντομα. Αν είχαμε, λένε οι άνθρωποι, ε, θέσεις εργασίας ε, και δημοκρατία, δεν θα φεύγει ο κόσμος. Είναι και μικρός ο πληθυσμός. Άρα και αυτό είναι μια ευκαιρία. Η πρόεδρος. Ναι. Όντω, μια τέτοια χώρα μπορεί γρήγορα να σταθεί στα πόδια τη αν έχει κανεί τα σωστά εργαλεία στα χέρια του. Βλέπω ότι και εσεί εδώ τι σημειώσει γιατί σα ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό και είστε συμπρόεδρο στην Επιτροπή ΤΕΚ. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατά σημειώσει για τα όσα διαμήθησαν για την Γκάμπια και τον όλο σχεδιασμό περί ανθεκτικότητας στην Γκάμπια πρέπει να βοηθάμε τις χώρες στη δημοκρατική τους μετάβαση για την οικονομική του σταθερότητα και όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ Τζιν για αυτήν την ενημέρωση. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το εκλογικό σύστημα. Λες βέβαια ότι λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κόσμος ήταν ε, πραγματικά πολύ σοκαρισμένος που δεν κοιτάμε τα δελτία ταυτότητας όσων ψηφίζουν. Ο καθένας έχει το δικό του ε, τρόπο να ψηφίζει. Δηλαδή αρκεί να ρίξει μια ματιά υπάλληλο αυτόν που έχει να ψηφίσει και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τέλο πάντων, ο καθένα έχει τι ιδιαιτερότητε του. Ευχαριστούμε, Τζιν. Um, Ευχαριστούμε, Τζιν, που ήρθε ω εδώ. Και να πάμε στο σημείο 7. να χειροκροτήσουμε την Τζιν και μετά να έρθουν ε, οι ειδικοί στο Προεδρείο. Okay, colleagues, now going to move on to... Συνάδελφοι, τώρα να περάσουμε στο σημείο 7. Διαχείριση φυσικών πόρων δασοκομείας. Διαφανής και βάση λογοδοσίας διαχείριση φυσικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες σε περίπτωση των δασών. Υπάρχει και link για την έκθεση που είχε καταρτιστεί από την Επιτροπή μας στην αποστολή στο Καμερούν. Ε, οι συνάδελφοι ευτυχώ είναι εδώ, ο κύριος Μαρσελέζη είναι εδώ λόγω χάρη και είχαμε ζητήσει έκτοτε μια μελέτη για τα νοσοκομεία για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί το να διαχειριζόμαστε του βασικού πόρου, το να του προστατεύουμε είναι σημαντικό όχι μόνο για την και μα πολιτική αλλά και για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ξέρουμε ότι πολλά πράγματα αλλάζουν και ότι αν δεν έχουμε βιώσιμη διαχείριση των δασών, αντίκτυπο θα υπάρχει μόνο όχι μόνο για τις ε, δασοφόρες χώρε αλλά και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Εδώ λοιπόν έχουμε την παρουσίαση της σχετικής έκθεσης. Την έχετε μπροστά σας. Έχω τον Πάτρικ Βέμς στα αριστερά μου, ο οποίος είναι σύμβουλος στην ΕΚΡΑΦ για θέματα δασοκομείας και ο κύριος Πίτερ Μίναν από τον ίδιο οργανισμό. Θα μας πείτε περισσότερα εσείς για τον οργανισμό σας και για τη δουλειά σας από την ΙΚΡΑΦ. Κύριε Βόλμφ, Παρουσιάστε μας την έκθεση. Δύσκολο το καθήκον. 70 σελίδες είναι η εκθέση. Πώς να τη συνοψίσω σε μια παρουσίαση που να σας αφήσει και κάποιες ε, βασικές ιδέες για το πώς γίνεται η διαχείριση των φυσικών πόρων στις χώρες αυτές. Ε, δύο λόγια πρώτα για το e-Craft, Διεθνές Κέντρο για την Έρευνα στην Αγροδασοπονία. Έχουμε την έδρα μας στον Ναϊρόμπι και θέλουμε να μελετήσουμε το ρόλο των δέντρων ε, στα τοπία. Να καταλάβουμε δηλαδή πώς τα ζώα, οι καλλιέργειες, οι άνθρωποι, τα ζώα μπορούν να αλληλεπιδρούν περισσότερο προς όφελος όλων. Βέβαια, η ρύθμιση των φυσικών πόρων έχει μεγάλη σημασία, ότι πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Άμεσο όφελος αφενός, ε, κόβοντας και πολλώντας κάτω και αυτό να το συνδυάσουμε με τη βιωσιμότητα των πόρων. Ε, στο πλαίσιο αυτό τα δάση πραγματικά είναι ένα σημαντικό θέμα. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να σας ε, παρουσιάσω τη μελέτη, το στόχο μας πρώτα απ' όλα. Αυτό που θέλουμε είναι να καταλάβουμε η λογοδοσία και η ευθύνη τι ρόλο διαδραματίζουν ε, στην ε, δασοπονία για τις ανθρώμενες χώρες που παίρνουν μεγάλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθήσαμε τον πιο κλασικό τρόπο, αναφέρουμε τη βιβλιογραφία και μετά κάνουμε μία μελέτη στο Καμερούν, την Κάνα και την Τανζανία. Και αυτοί που πήγαν στο Καμερούν φαντάζομαι θα μπορούν να μας ε, ε, κάνουν τις ερωτήσεις τους. Διαλέξαμε αυτές τις χώρες που είναι σε διαφορετικά στάδια συμμετοχή στο ΦΛΕΚΤ και κάθε μία χώρα καλύπτει ε, μία από τις τρεις βασικές δασικές περιοχές της Αφρικής. Έτσι έχουμε πολλές και διαφορετικές πληροφορίες. Πριν έρθω στις λεπτομέρειες, να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη η πυκνότητα του πληθυσμού, το ίδιο και τα δέντρα στην Αφρική. Άρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατάχρησης ε, για ε, βραχυπρόθεσμο όφελος από τους Αφρικανούς. Αλλά καλύτερα να το χρησιμοποιούν για μακροπρόθεσμο όφελος, ε, που θα ήταν ε, το δάσος ενώ οι Αφρικανοί. Λοιπόν, το πάραν. κοιτάμε το νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση πληροφορίε, για την ενθάρρυνση, μια συζήτηση που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, δημόσια ευθύνη και λογοδοσία των διαφόρων φορέων, να δούμε αν ήταν ε, έγκαιρη πληροφόρηση, αν ήταν εύληπτη κτλ. κτλ. Διαφάνεια στις ε, παραχωρήσεις, ε, εκχώρηση δικαιωμάτων, ήταν θέματα που μας απασχόλησαν και βέβαια ακόμα πιο σημαντικό διαχείριση εσόδων. Σημαντικό να δούμε και του εποπτικού μηχανισμούς, τους μηχανισμούς λογοδοσίας, αν είναι αποτελεσματικοί. Και επίσης θα πρέπει να καταλαβαίνουν και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς το τι γίνεται. Διαφάνεια λογοδοσία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι σημαίνει όμως διαφάνεια τελικά. Σημαίνει επικαιροποιημένα ακριβή δεδομένα, πλήρη δεδομένα που θα πρέπει να είναι και προσαρμοσμένα στι ε, απαιτήσει και στι ανάγκε των διαφόρων χρηστών. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν και μια διεθνή μελέτη. Αυτοί μπορούν να θέλουν κάτι τελείω διαφορετικό από τι τοπικέ κοινωνίε που έχουν πάει σχολείο τα μέλη του για λίγα χρόνια μόνο. Θα πρέπει επίση να τα δούμε αυτά, τη διαχείριση των πόρων, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση των προγραμμάτων. Το σλόγγαν δηλαδή είναι οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, και ίσω είναι και τα πιο δύσκολα που πρέπει να πετύχουμε. Τώρα η λόγοδο έχει να κάνει με την αξιοπιστία τη διαδικασία για την παρακολούθηση, τη διαδικασία εκχώρηση δικαιωμάτων και έσπραξη εσόδων. Μηχανισμοί υποβολή αναφορών. Στην πράξη λειτουργούν, στη θεωρία είναι καλοί αυτοί οι μηχανισμοί, μπορούν να βελτιωθούν κτλ. κτλ. Συνεχώ πρέπει η συλλογή ε, και η μέθοδο ε, να βελτιώνονται και αυτό σε όλα τα επίπεδα. Πριν πάω στι λεπτομέρειε μελέτη, δυστυχώ πρέπει να σα πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι οι τάσει είναι ανησυχητικέ στην αγροπονία. Επειδή δεν μπορείτε να το διαβάσετε αυτό, το έχουμε μετατρέψει σε ένα πίνακα λίγο καλύτερα, καλύτερο από το προηγούμενο. Βλέπετε την ε, μπλε γραμμή και βλέπετε ότι μειώνεται και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ε, η κόκκινη γραμμή που μειώνεται, τα αρχαίγωνα δάση. Βλέπετε και την πράσινη γραμμή, η οποία από το 2000, και ούτε και εγώ το διαβάζω από εδώ, τι γίνεται με το ΤΙΚ ε, και τα λοιπά. Για να δούμε τα πορίσμα της μελέτης. Τα βασικά. Η θολωτική συμφωνία φλέκτα και η κανονασμός για την ξυλία είναι τα βασικά μέσα που επηρεάζουν και τα οποία πρέπει να λεπιδρούν τα την δασοπονία. Το έχει δείξει και η βιβλιογραφία, όχι μόνο για τις χώρες που μελετήσαμε, αλλά παγκόσμια βιβλιογραφία. Είναι αρκετό το ποσό που έχει επενδυθεί ε, στο ΦΛΕΚΤΑ, 200 εκατομμύρια ευρώ και σε σχετικές δραστηριότητες ε, και είναι θετικός αντικτύπωση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη διακυβέρνηση. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε αυτά κονδύλια, να καταπολεμήσουμε την παράνομη λοτομία, να βελτιώσουμε τη διαχείριση των δασικών πόρων και να στηρίξουμε τι ε, κυβερνήσει και διοικήσει των κρατών για τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των συμφωνιών με του διάφορου εμπλεκόμενου φορεί. Πού πάνε αυτοί οι πόροι λοιπόν τη Ένωση, πρώτα απ' όλα στην πληροφόρηση, νομικέ μεταρρυθμίσει, στην διαφάνεια, που είναι και ε, η βάση για τη χρηστή διακυβέρνηση. Σε επίσης ε, θέματα που έχουν να κάνουν ε, με την παρακολούθηση και την τη νησιότητα. Και το τρίτο είναι οι εγχώριες αγορές. Εδώ πάλι δεν βλέπετε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Θα σας πω τι λέει λέει που έχουν πάει τα χρήματα αναχώρα χώρα και ανατομέα. Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση για περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ βλέπετε κάτι πιο εύληπτο, ευτυχώς, δηλαδή 7 χαρακτηριστικά του τομέα αυτού, στην Αφρική πάντα. Το πρώτο είναι τα νομικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την χάραξη πολιτικής με βάση επιστημονικά δεδομένα, λογοδοσία και χάραξη πολιτικής ή ε, πληροφόρηση. Τι βλέπουμε, Στη Λιβερία το 2010 πέρασε ένας νόμος για την ελευθερία πληροφοριών, αλλά 7 χρόνια μετά βλέπουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί παρά με πολύ αργούς ρυθμούς. Τανζανία και Γκάνα έχουν νομοθεσία για την ελευθερία αυτή της πληροφορίας, θεωρητικά όμως, γιατί δεν υπάρχει σχετικός νόμος. Το ίδιο για Καμερούν και Κονγκό δεν υπάρχει καν δηλαδή, νομοθεσία εκεί. Και επίσης ε, δεν υπάρχει καν ευαισθητοποίηση για το ρόλο που θα είχε ένα τέτοιο νομοσχέδιο στην Ουγγάντα. Λάβω σκουμπιπάτσα, Δεύτερο χαρακτηριστικό, ποιότητα, εγκαιρότητα, προσβασιμότητα των πληροφοριών ε, στο κοινό. Πάλι ποικίλουν ε, αυτά που είδαμε στις διάφορες χώρες, παραδείγματος στο Καμερούν. Υπάρχει ε, πρόσβαση ελεύθερη σε ένα αποθετήριο, online reposter όπως λέγεται. Πρακτικά βέβαια περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για να βασίσουν εκεί τις αποφάσεις τους. Στη Λιβυρία η κατάσταση είναι καλύτερη υποτνέει ότι υπάρχουν πληροφορίε για τις δραστηριότητες, τα διαχειριστικά σχέδια, την κατάσταση των δασικών πόρων. Είναι δημόσια με αυτά τα στοιχεία. Ουγγάντα, Γκάνα, Τανζανία. Θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά πολύ λίγο είναι τι πληροφορίε. Τώρα, διαφάνεια σε ό,τι αφορά παραχωρήσει και εκχώρηση δικαιωμάτων. Κονγκό Μοζαμβίκη έχουν νομικά εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ε, πληροφορίες που αφορούν τις εκχωρήσεις. Καμερού, Τανζανία, Γκάνα ούτε ενημέρωση έχουν ούτε διαφάνεια για τι άδειε και για τις εκχωρήσει. Άρα δύσκολα καταλάβει κανεί τι συμβαίνει και στη κεντροαφρικανική δημοκρατία υπάρχει υποχρέωση να ενημερώνονται οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς. Αλλά δεν γίνεται και πράξη. Σε ό,τι αφορά διαχείριση εσόδων, Ανιγυρία, Αγκόλα, Κονγκό δημοσιεύουν πληροφορίες ε, χρηματοπιστωτικές πληροφορίες και ε, άλλα που έχουμε κάνει μέσω. Δεν κάνω τανζανία, πηγαίνουν τα χρήματα στα δημόσια ταμεία, άρα η διαφάνεια είναι λιγότερη, αν δεν ξέρει κανείς ε, πώς πάνε αυτά τα χρήματα μετά. Όταν μιλάμε για επιπτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης, Καμερούν, Κογκό, Λιβύρια έχουν ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς, η Τανζανία όχι. Και Όταν μιλάμε για τους μηχανισμούς λογοδοσίας, εδώ ε, τα πράγματα είναι παρόμοια σε όλες τις χώρες. Περιορισμένη πληροφόρηση για την ευστερική λογοδοσία. Τέλος. Τι γίνεται με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των, ε, της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες χώρες έχουν κάποιους κανόνες σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση για τη διαφάνεια και την λογοδοσία. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς, εδώ τι βλέπουμε. Δύο πράγματα. Πρώτον, αυτοί οι φορείς, μηχανισμοί, θελοντικές συμφωνίες, red scene, θα έπρεπε να αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη, αλλά είναι πρωτοβουλίε ξεχωριστέ. Δεν υπάρχει επικοινωνία ούτε σχέση εργασία. Το ίδιο έχουμε και με την αναπτυξιακή βοήθεια στη περιοχή. Δηλαδή υπάρχει προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των project, αλλά στην πράξη αυτό καθίσταται ιδιαίτερω δύσκολο. Επίση, πολύ λίγα στοιχεία στηρίζουν την υπόθεση ότι οι εθελοντικέ συμφωνίε δίνουν κίνητρα για την ε, βιώσιμη διαχείριση επιτόπου, δηλαδή με το να προσελκύουν νέου συμμετέχοντες στο μηχανισμό FLECT. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές νόμιμης ξυλίας χάρη στα μέτρα αυτά. Όχι βέβαια σε μεγάλο βαθμό. Ποιε είναι τώρα οι βασικέ προκλήσει. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει ανάπτυξη στην αγορά, αλλά πολύ λιγότερο αφορά την Ευρώπη. Έχουμε μεγάλη αύξηση της εγχώριας ζήτησης και από αγορές αναδιόμενες όπως η Κίνα. Δεύτερον, είναι αφανής ή θα αν θέλετε παράνομη, επειδή είναι μικρής ε, κλίμακας και βιοτεχνική η βιομηχανία αυτή. και εκπροσωπεί πάνω από το 70% σε χώρες όπως το Καμερού και η Γκάνα. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις, ευθύνονται για τη μεγάλη πλειοψηφία ε, της παράνομης υλοτομίας. Ποιες είναι οι συστάσεις μας για την Κομισιόν, και ε, για την Επιτροπή σας. Πρώτον, καλό θα ήταν ορισμός της νομιμότητας ε, να επεκταθεί και να περιλαμβάνει στο δυνατόν ευρύτερη δέσμη ασφαλιστικών δικλείδων για τα δικαιώματα και τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Δεύτερον, καλό θα ήταν ε, να, μιλήσει κανείς σε μεγάλες αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Κίνα, για να μπορέσουν αυτές οι χώρες να θετήσουν παρόμοια πρότυπα με το ΦΛΕΚΤ για τις δικές τους εισαγωγές αφρικανικού ψήλου. Τρίτον, Χρήσιμο θα ήταν να εστιάσει και η προσοχή και η επένδυση και οι δράση εσωτερικέ, εσωτερικές αγορέ αγορές ε, ξυλίας, ιδίως από μικρούς ε, ε, επιχειρηματίες. Τέταρτον, θα πρέπει να υπάρξει δημιουργία δαμών πέρα από την παρακολούθηση, την ανίχνευση και την εποπτεία. Θα πρέπει επίση να υπάρχουν συνέργειε μεταξύ των διαφόρων εργαλείων και αυτό μπορεί να το ε, επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι δράσει τη, τέλο θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι κίνητρα θα μπορούσαμε να δώσουμε για την βιώσιμη διαχείριση ε, στην Αφρική και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάω πάντα για τους μικρούς ε, ε επιχειρηματίες, το premium pricing και το labeling είναι σημαντικά στοιχεία. Βέβαια θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τα πράγματα, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε πολλή ενημέρωση για το πλήρε κόστο και όφελο από την Θελοντική Συμφωνία από το e UTR. Μέχρι στιγμή αυτέ οι διαδικασίε ε, ε, χρηματοδοτούνται από τα δημόσια οικονομικά και λίγε είναι αξιολογήσει ε, σε ό,τι αφορά το πλήρε κόστο αδειοδότηση, της αγωνιστικότητας του αδειοδοτημένου ξύλου κτλ. Δεν είναι προκλήσει αλλά είναι και ευκαιρίε. Παραδείγματο χάρη, μεγαλύτερη παρακολούθηση για του στόχου ΑΙΤΣΙ και για τους ε, βιώσιμους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, ε, έχουμε τη δήλωση της Νέας Υόρκης για τα δάση. Θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα ε, σε σχέση με αυτή τη δήλωση και να έχουμε συμπεφωνημένους στόχους και να χρηματοδοτούμε βάση επιδόσεων. Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη λογοδοσία και την διαφάνεια για τις δραστηριότητες των Αφρικανικών μελών και επίσης θα μπορούσαμε να προωθήσουμε συμπράξεις δημόσιο ειδικού τομέα και θα ολοκληρώσω με τρεις ε, ε, διαφάνειες με μια μελέτη περίπτωση για την Κάνα. Η Κάνα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία απευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υλοτομία πριν μάλλον ξεκινήσει ε, η εξόριξη πετρελαίου. Ω εκ τούτου έχει χάσει 34% των δασών τη από τη δεκαετία του 1990. Αποφάσισε η χώρα αυτή να υιοθετήσει το μηχανισμό φλέκτη για να έχει ε, συνεχόμενη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 60% της ολοτομίας, ε, των προϊόντων ολοτομίας πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά είναι και ένας μηχανισμός ε, της κυβέρνησης για να μεταρρυθμίσει έναν απορριθμισμένο στο παρελθόν τομέα. Οπότε ξεκίνησε τη διαδικασία το 2009, επικυρώθηκε το 2010 και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα ξεκινήσει τώρα σύντομα τι επιλογές υπάρχουν για ευρωπαϊκή ενίσχυση. Να διερευνήσουμε κατά το δυνατόν την μικρή κλίμακα σελοτομία. Γιατί στην Κάνα ε, το 80% της εσωτερικής ε, ξυλίας αλλά και αυτής που εξάγεται ε, προκύπτει από εκεί και απασχολεί περίπου 138.000 άτομα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την ε, κυβέρνηση να δώσει τέτοιες νόμιμες ε, διεξόδους για τους ε, μικρούς λετόμους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα νομικό καθεστώς, να υπάρχουν μηχανισμοί και εργαλεία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες και προϋποθέσεις, τεχνική στήριξη, να μεταδίδεται δηλαδή εμπειρία από άλλες χώρες που υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα και να υπάρχει και μηχανισμός διαβούλευσης και φόρα ε, για να λαμβάνονται υπόψη οι προβληματισμοί και ανησυχίες αυτών των ε, μικρών υλοτόμων. Αυτά είναι ο λίγης από εμένα. Είμαι στη διάθεσή για τυχόν Okay, thank you very Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το, λόγο στον κύριο Μάρσελ Λέσλι που ε, δεν ξέρω, θέλετε να μιλήσετε απευθεία γι' αυτό ή να μας πείτε για την αποστολή και τα πορίσματά σας. Έχουμε αυτές τις επιμέρους ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, BA ε, και FLECT. Ε, τι πρέπει να έχουμε εμείς ε, κατά νου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο μηχανισμών, η κατάσταση επιτόπου αντιμετωπίζει το ένα και το άλλο τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Δώστε μας μερικά στοιχεία γιατί δεν είμαστε και όλοι ειδικοί σε αυτά τα θέματα. και η νομοθεσία FLECT ε, εξετάζεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας παρουσιάσω τα της αποστολής στο Καμερούν, 22 με 24 Μαΐου. Ε, ήμασταν οι βουλευτές, ο κύριος Έγκελ, ο κύριος Αγγιλάρ και εγώ ίδιος, ο κύριος Σρέντερ από την Επιτροπή Ανάπτυξης και η συντονίστρια των Πρασίνων. Είδαμε πάρα πολλούς μέσα σε τρεις μέρες εκπροσώπους θεσμικούς της, πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρηματιών και άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα. Ευχαριστώ την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί για την δουλειά τους και την υποδοχή τους. Πολύ χρήσιμα για να δούμε τα θέματα ενδελεχώς. Εντάχει η διάγνωση για να περάσω αμέσω στις συστάσεις. Γιατί έγινε αυτή η αποστολή. Γιατί είδαμε κάποια πράγματα και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ε, παράγοντας μόχλευσης για να βοηθηθούν κάποιες καταστάσεις. Η βασική ερώτηση ήταν αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι το φλεκτ στο Καμερούν. Η ερώτηση και η απάντηση που εμείς δώσαμε ως ε, αντιπροσωπεία ήταν ότι ναι, να συνεχιστεί το φλεκτ, αλλά να τεθούν επιτάπητος και κάποια ουσιώδη ζητήματα, ώστε το φλεκτ να έχει πραγματικό όφελος ε, για τη χώρα. Να επενθυμίσω τι ημερομηνίε εδώ για την εταιρική, τη Συμφωνία Εταιρική ε, σχέση που άρχισε να ισχύει από το 2008 μέχρι τις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018, με συγχωρείτε, δεκαετής ε, διάρκεια και στο τέλος της εταιρικής σχέσης τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν αν θα θέσουν επιτάπητος κάποια θέματα ή αν θα υπάρξει παράταση και ανανέωση της συμφωνίας ε, χωρίς να συζητηθεί. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα παριθμίσω και μας φαίνονται σημαντικά για τη συνέχεια των εξελίξεων. Πρώτον, ό,τι έχει να κάνει με τη κυβέρνηση, την διαφάνεια και την διαφθορά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, ε, το πιο έτσι ογκώδες που απασχόλησε Διακυβέρνηση, διαφάνεια και διαφθορά λοιπόν συζητήθηκαν και είδαμε ότι υπάρχει διαφορά ως την υλοποίηση του ΦΛΕΚΤ στο Καμερούν για έναν βασικό και γνωστό λόγο που είναι η ε, απομόνωση. Η απομόνωση των Υπουργείων μεταξύ τους. Δεν συνεννοούνται. Ο καθένας τα κάνει όπως θέλει. Αλλιώς θα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλιώς ε, της Χορταξίας, αλλιώς ε, της Γεωργίας. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ε, η πραγματική υλοποίηση της εταιρικής σχέσης προ το ΦΛΕΚΤ. Έπειτα για την ε, εφαρμογή των νόμων. Στο Καμερούν είδαμε ότι νόμοι υπάρχουν. Δεν είναι και το πρόβλημα. Νόμοι εγκρίνονται. Υπάρχει ένα καλό πλουστάσιο. Αυτό που δεν υπάρχει όμω είναι η πραγματική εφαρμογή των νόμων στην πράξη. Και επιπλέον αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι στην περίπτωση τη εταιρική σχέση υπάρχει ένα δίχτυο νομιμότητα για να φτάσει κανείς να αποστοποιήσει το, τα προϊόντα υλοτομίας, αλλά είναι πραγματικά περίπλοκο για να υπάρχουν τα πιστοποιητικά. Είναι λοιπόν σημαντικό για να βγουν τα πιστοποιητικά να υπάρξει απλούστευση και επίσης για να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Διότι όσο πιο περίπλοκο είναι το σύστημα, σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο μπορεί να υπάρξει διαφθορά. Ένα σημαντικό πράγμα και επειδή μιλάμε για νόμους... Για να ολοκληρωθεί το νομοθετικό οπλοστάσιο, κυρίω οι νόμοι περί δασοκομεία που θα πρέπει να υλοποιηθούν, είναι σημαντικό να υπάρξει και αυτή η πραγματική εφαρμογή. Για τι συστάσει τώρα. Υπάρχει ένα ιστότοπο ε, με πληροφορίε για να μπορεί κανεί να παρακολουθήσει την κατάσταση των δασών. Ήταν επί μήνε μη διαθέσιμο πρόσφατα ξαναοργανώθηκε και δεν είναι καθόλου επικαιροποιημένο. Υπάρχει λοιπόν πρόσβαση στο ίντερνετ σε αυτές τις πληροφορίες, αλλά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Και κάτι που μου φαίνεται επίση σημαντικό, που ακούστηκε και πριν, είναι ο συντονισμό. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών προγραμμάτων, δηλαδή φλεκτ και RECT ε, προκειμένου. Οι στόχοι είναι αρκετά παρόμοιοι, μιλάμε για δάση. Και όμως δεν υπάρχει απαραίτητο συντονισμός για να υπάρξει δραστική παρέμβαση. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο συντονισμός και η ολοκλήρωση, η συμπερίληψη της ξυλίας, της διαδικασίες διαφάνειας για τις εξωτερικές ε, βιομηχανίες, κάτι που ισχύει και για τα κλιβερία λόγου χάρη. Πρέπει να το κάνουμε και στο Καμερούν. Επίσης, μια και μιλάμε για κυβέρνηση και διαφάνεια, αυτή τη στιγμή το Καμερούν ολοκληρώνει το σύστημα πληροφορίας για τους δασικούς πόρους, το ΣΥΖΙΦ. Ε, αλλά υπάρχουν διαρκώ φραγμοί σε αυτό το σύστημα πληροφορία και την διοργάνωσή του. Έχει μπλοκαριστεί η διαδικασία και ελπίζουμε τον Οκτώβριο να έχει τελειώσει. Σύστασή μα όμω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επαφείται μόνο στο ΣΥΖΙΦ. Ε, ελπίζουμε να υπάρχουν και άλλοι πόροι για να ενημερωθούμε από ότι το ΣΥΖΙΦ. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών Υπήρχε μια θετική διάσταση στο Καμερούν ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμμετάσχει και να έχει φωνή, να κάνει τη φωνή της να ακουστεί. Αυτό επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ακούσει την κοινωνία των πολιτών που ήταν διαρκώς παρούσα στην όλη διαδικασία. Ήταν παρούσα όμως δεν ήταν παρούσα στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Ενώ ήταν παρούσα μάλλον στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, ε, δεν ήταν το ίδιο στην ε, πραγματική υλοποίηση της εταιρικής σχέσης και μετά στην ε, παρακολούθηση του πώς προχώρησε η εταιρική σχέση. Εκεί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από του εταίρους τη στο Καμερούν να εξασφαλίσουν την παρουσία τη κοινωνία των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. στην αρχή, τη μέση και το τέλο. Επίσης, η αποστολή εξωτερικών παρατηρητών. Δεν υπάρχουν πια. Όλοι οι εξωτερικοί φορείς οι ανεξάρτητοι φορεί ε, λείπουν, το είπαν οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών, πρέπει να είναι εκεί για να μπορούν να δουν τι προσφέρεται μέσω τη εταιρική σχέση και το ΦΛΕΚΤ. Και να υπάρχει πιστοποίηση τη ξυλία με σαφεί προδιαγραφέ. Επίση, για μια σύσταση που μα κάνατε και πρέπει να μεταφερθεί σε Βίκο ΑΟΤΑ, είναι η κοινότητα των εμπειρογνωμόνων, όχι μόνο για το Καμερούν, αλλά σε όλη την περιοχή του κόλπου του Κονγκό, της Λετάνης του Κονγκό, για να υπάρχει μια σαφής ε, έποψη του τι συμβαίνει. Και να ε, μπορούν οι παρατηρητές να μας ενημερώνουν. Ο λόγου Χαριοκόφη Ενάν θα μπορούσε να είναι επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας για να παρακολουθεί την υλοποίηση του ΦΛΕΚΤ στην όλη περιοχή το δεύτερο σε έκταση τροπικό δάσος του κόσμου. Και το άλλο που πρέπει να προσθέσω και να είμαστε σαφείς ως προς αυτό είναι ότι το φλεκτ δεν μπορεί να είναι απομονωμένο αλλά και το πρόγραμμα για την ε, υλοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή το ΦΛΕΚΤ είναι σημαντικό για τον Νότο, αλλά και τα ε, δασοκομεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πρέπει να υλοποιούνται σωστά. Και τρία σημεία έχω να παρατηρήσω εδώ. Πρώτον, θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη δεν αφοσιώνουν του απαραίτητου ε, ανθρώπινου και τεχνικού πόρου, ώστε οι αρμόδιε αρχέ να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Κάποιοι ναι, βέβαια, το είδαμε στι κάτω χώρε. Αλλά το Βέλγιο λόγου χάρη είναι το πρώτο σημείο εισόδου τη ξυλία από το Καμερούν και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο εργάζεται ε, σε απασχόληση μερικής, μερικού χρόνου. Ε, δεν έχει καμία πραγματική ε, ειδική γνώση για τη δουλειά του. Επιτά πρέπει να υπάρχουν κυρώσει, γιατί γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρο τη ξυλία των προϊόντων υλοτομία που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράνομα, είναι υψηλό κινδύνου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν πραγματικέ κυρώσει. Οι κάτω χώρε επέβαλαν κυρώσει, άλλε χώρε όμω δεν το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση να χρησιμοποιείτε το δίκαιο περί ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για αυτά όσα έρχονται απ' έξω προ τα μέσα. Και επίση κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Τελευταία παρατήρηση, επίση ε, ιδιαίτερη σημασία, κάτι που είναι εντελώ ε, θαλμοφανέ για όλου του παραγόντε, είναι η Κίνα. Δεν μπορεί τίποτα να γίνει αν οι Κινέζοι δεν συμμετάσχουν. Οι Κινέζοι ξέρουμε ότι έχουν αυτή την οριζόντια προσέγγιση στα πράγματα που δεν ε, χρησιμοποιεί κανένα κριτήριο ποιότητα, κανένα κριτήριο κοινωνική δικαιοσύνη, κανένα κριτήριο. Θα μπορούσα να συνεχίσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τι γυναίκε και το καθεξή. Θα μπορούσα λοιπόν να, να μιλάω για ώρε γι' αυτό, αλλά έχουμε πραγματικό πρόβλημα με την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι ώστε να έχει ένα σοβαρό σύμμαχο για την καταπολέμηση τη αποψήλωση και τη παράνομη φιλοτομία. Τέλο, για να ολοκληρώσω πολύ γρήγορα κάτι που επανήλθε ε, επανειλημμένο στι συζητήσει μα το δικαίωμα των ηθαγεν... Τα δικαιώματα των ηθαγενών, ένα θέμα όπου δεν έχουμε κάποια λύση του προβλήματος. Υπάρχουν πολλοί νόμοι, αλλά το δίκαιο των ηθαγενών και η προστασία των δασών, πολύ περίπλοκη κατάσταση. Είναι περίπλοκο να καταλάβει κανείς ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν ηθαγενείς, λέει, οι οποίοι απειλούνται πραγματικά από την αποψήλωση των δασών και ένα από τα σημεία που επίση εφήγει πάρα πολύ στι συζητήσει μα και που εμένα με απασχόλησε ιδιαίτερω για την εξακολούθηση και τη συνέχεια των εξελίξεων στο Καμερούν είναι το μοντέλο ανάπτυξη που θα χρησιμοποιήσει το Καμερούν ω το 2035, που βασίζεται στην γεωργική βιομηχανία, στι μεγάλε εκμεταλλεύσει. Χρειάζεται, όπω είπαμε, να προστατευτούν και οι μικρέ εκμεταλλεύσει. Το Καμερούν όμω έχει επιλέξει το αντίθετο στο μοντέλο ανάπτυξή του και το λέει. Το, ε, οι μεγάλε εταιρείε, οι μόνο καλλιέργειε θα μας επιτρέψουν να ξεφύγουμε από την ε, χαμηλή ανάπτυξη, τη μηδενική ανάπτυξη που θεωρούν ότι έχουν. Εμείς νομίζουμε ότι αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Αφρονούμε ότι πρέπει να μπει στο κέντρο της συζήτησης η, η όλη μετατροπή, μετατροπή των γεών ε, των δασών σε μονοκαλλιέργειες για την καλλιέργεια καουτσού, καφέ και άλλων. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς το ΦΛΕΚΤ μπορεί να ε, συμβαδίσει με το αναπτυξιακό μοντέλο του Καμερούν και τη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Μια σημαντική υπηρεμενία που φτάνει το 15 Δεκεμβρίου 2017, τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει επιτάπητο στα γεωγραφικά αυτά θέματα και να αποφασίσει μαζί με τον εταίρο τη εάν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Επίση, πρέπει να του ζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα προβλέψουν στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων για να μπορέσουμε να είμαστε επικοδομητικοί στην προσέγγιση μα στο Καμερούν και γύρω-γύρω. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ε, ιδιαίτερα ευαισθητομένη επισκόπηση. Έχει καιρό να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα. Είχαμε την, ε, τον κανονισμό για την ε, υλοτομία, μετά είχαμε το FLEC-TPA. Πρέπει να έχουμε αρχικά μια καλή εικόνα για το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα. Έχουμε ένα σύστημα διαπίστευσης Εξετάζουμε διάφορα προγράμματα λοιπόν και είναι πολύ περίπλοκα. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακριβώ πώ ε, λειτουργούν στην πράξη. Είπατε ότι υπάρχουν μελέτε για τον αντίκτυπο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Επιτροπή πάντα βεβαίω κάνει αξιολόγηση ε, των εργασιών τη, αλλά θέλαμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό και για την Κίνα. Δεν ξέρω κατά πώς υπάρχει ε, συζήτηση, υπάρχουν επαφέ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα για να μπει και Κίνα σε αυτέ τι διευθετήσει. Ιδάλω, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, δεν βλέπουμε ότι πώς μπορεί να υπάρξει η λύση. Δηλαδή, αν απλώς ε, ε, περάσει η ξυλία, η η δραστηριότητα από την Ευρώπη στην Κίνα, τότε το πρόβλημα παραμένει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μινάγκ. Πολύ χρήσιμε οι παρατηρήσει σα. Ξεκινώ από τις διαδικασίε Black TPA και EUTI. E ε, το δεύτερο καθεστώς ε, είναι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι για ο εισαγωγής ξυλίας ε, υποχρεούνται ε, να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια και να αποδεικνύουν ότι η ξυλή αυτή είναι νόμιμη και από διαπιστευμένες πηγές. Όπως ανέφερε και ο κύριος Μασιλεσί ε, προηγουμένως, υπάρχουν τεράστια ζητήματα από πλευράς λογοδοσίας ε, και στην Ευρώπη, αλλά και από πλευράς οικοδόμησης δυνατοτήτων, γιατί δεν υπάρχει επαρκής δεν υπάρχουν υπαρκείς δομέ για να διεξάγονται αυτέ οι ε, διαδικασίες. Έτσι ξεκίνησαν όλα αυτά το 2013. Στην νότια πλευρά, αν θέλετε, έχουμε τη διαδικασία FLECT VPA. Το FLECT έχει τέσσερα βασικά ε, στοιχεία. Πρώτον, ορισμό ορισμός της νομιμότητας, της νόμιμας που εξαρτάται από την κάθε χώρα. Μετά, διασφάλιση ποιότητα και συστήματα διασφάλισης ποιότητα και μετά έχουμε τις ε, εθελοντικές εταιρικέ σχέσεις, όπου οι χώρες ε, εθελοντικά επισέρχονται και έχουν, ε, την έχουν προσυπογράψει αυτή. Και μετά έχουμε κατευθείαν γραμμές για την παρακολούθηση. Πώς δυσφαλίζουμε δηλαδή ότι η ξυλία όντως προέρχεται από τις σωστές νόμιμες πηγές. Οπότε εμεί περισσότερο, εστιάζουμε την προσοχή μα στην ε, αναπτυξιακή πλευρά, πλευρά δηλαδή Αφρική, παρά ε, στην ευρωπαϊκή διάσταση. Το είπε και ο κ. ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να λειτουργεί αμφίδρομα. Η μία πλευρά είναι να ελέγχουμε ότι όντω ασκείται δέωση επιμέλεια και στην, ε, κατά την εισαγωγή, αλλά και από την πηγή. Ξέρουμε ότι έχουμε τους κανονισμούς. Στις περισσότερες αυτέ τι χώρε οι νόμοι είναι εξαιρετικά περιπλοκοί, ε, αλλά υπάρχουν και δυνατότητε να παρακαμφθούν αυτοί οι νόμοι. Χρειάζεται λοιπόν και ιδέως επιμέλεια από την άλλη πλευρά για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αλλιώς ε, δεν έχει νόημα η όλη διαδικασία ή ε, εφαρμόζεται αναποτελεσματικά. Εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα της Κίνας όπως αναφέρατε και προηγουμένως. Αν δείτε τα γεωγραφικά στοιχεία ε, της ξυλίας και στην Ασία, θα καταλάβετε ότι δεν έχουμε να κάνουμε εδώ μόνο με την Κίνα, έχουμε δύο σημαντικούς ε, φορείς και το Βιετνάμ και η Μαλαισία έχουν μπει σε αυτό το χώρο. Πολύ συχνά αυτές οι τρεις χώρες δημιουργούν ένα περίπλοκο ε, δίκτυο εισαγωγής ξυλίας από το Λάσο, από την Καμπότζη και είναι δύσκολο κανείς να ανοιχνεύσει από πού προήλθε αυτή η ξυλία. Όταν λοιπόν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις συζητήσεις με την Κίνα, καλό είναι να το εξετάσει πιο ολιστικά. Γιατί το, οι επιχειρήσεις από το Βιετνάμ και τη Μαλαισία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες και αλεξαρτώμενες από κινέζικα συμφέροντα. Το Βιετνάμ αναπτύσσεται πιο γρήγορα από ε, την Κίνα, στην Κάνα, από, από άποψης ε, εισαγωγών. Και εδώ το σημαντικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα μιλάει για την ε, δασονομική ξυλία, την νόμιμη ξυλία που δίνεται ε, μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Τώρα όμως βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο εξηλία προέρχεται από μη δασονομικές ε, ε, πηγές, από φυτίες ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί στην Αφρική πολλή ξυλία αφήνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όταν καθαρίζονται οι ε, φυτίες κακάο. Και επειδή απέχουν πολύ από τις πόλεις και από τα δικά δίκτυα, πολλή ξυλία προκύπτει από τις εκμεταλλεύσεις, γιατί είναι πιο φτηνό να τις ε, μεταφέρουμε από ε, τις εκμεταλλεύσεις προς την πόλη και είναι η ίδια η ποιότητα του ξύλου, η ίδια ηλικία και σκληρό πολύτιμο ξύλο κατά βάση. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι θα κάνει με αυτή την ε, μη δασονομική ξυλία από τις φυτίες και από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί είναι το 90% της εσωτερικής εκμετάλλευσης, ε, της κατανάλωσης συγγνώμη, του Καμερούν και ίσως είναι πάνω από 30% των εξαγωγών, εκτιμούμε εμείς, τα τελευταία χρόνια. Πολύ από την ξύλια που πάει στο Βιετνάμ από την Κάνα δεν είναι από τα δάση, είναι από τις εκμεταλλεύσεις. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε σε ένα αγροτασνομικό πλαίσιο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το μέλλον ε, της ξυλίας ε, στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Αν δείτε την ακτή του Ελεφαντοστού, την Γκάνα, πολλοί από αυτή την ξυλία δεν προέρχεται από τα δάση, δεν έχουν πλέον δάση σχεδόν. Από πλευράς πολιτικής λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε ευρύτερα αυτό το σημείο και να δούμε και άλλες επιλογές, που μπορούμε να το, να το συνδυάσουμε το FLECT με άλλες, άλλους τομείς πολιτικής και πρωτοβουλίας. Στο επίκεντρο έχουμε τις αφρικανικές ε, χώρες. Αντίστοιχα έχουμε και χώρες που ε, εμπλέκουν τεράστιες εκτάσεις ε, στο Red Plus. Με πολύ φιλόδοξες ε, πολιτικές δίνουν χώρα σε τεράστιες επιχειρήσεις που ανοίγουν γεωρικές εκμεταλλεύσεις για διάφορες καλλιέργειες. Αυτή η πολιτική από το Υπουργείο Γεωργίας αφαιρεί τεράστιες εκτάσεις από ό,τι αυτές που έχουν δεσμευθεί υπό το Red Plus και τις ευρύτερε πολιτικές του ΟΗΕ για την μείωση των εκπομπών. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν μερικά βασικά μηνύματα. Πρώτον, πρέπει αυτές οι χώρες να πάρουν αυτό το θέμα στα σοβαρά από πλευρά διακυβέρνηση, όπω είπε και ο κ. Μασελίση, πώ όλα αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη. Γιατί υπάρχει το νομικό πλαίσιο, πλαίσιο υπάρχουν τα συστήματα, αλλά δεν εφαρμόζονται συνήθω. Δεύτερον, πρέπει να το εξετάσουμε ευρύτερα το θέμα, όχι μόνο σε φλεκτ, γιατί έχουμε και Κίνα, Βιετνάμ, Μαλαισία, ε, που είναι σημαντικοί παίκτε, μπαίνουν στο χώρο και εξουδετερώνουν ενδεχομένω οτιδήποτε μπορεί να μας φέρει το φλεκτ σε 5-10 χρόνια. Και μετά πρέπει να δούμε τι σημαίνει με την ξυλία πέραν των δασών οι εκμεταλλεύσει και φυτίες σημαντικό φορέας ξυλία και όλο και περισσότερο αποτελούν πηγή παράνομης υλοτομήσης. Ε, που, και αυτή η ξυλία έρχεται στην Ευρώπη αλλά πάει και στην Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε και μια συζήτηση στην Ολομέλεια για, για την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το πάνελ υψηλού επίπεδου για του ε, στόχους βιώσιμη ανάπτυξης στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο και έχουμε συμφωνήσει πρόσφατα και για την αντιστοιχική πολιτική. Όμως όλα αυτά συνδέονται με τις εσωτερικέ πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέτε ουσιαστικά ότι τα όσα κάνουμε για τη Συμφωνία των Παρισίων θα πρέπει να αντιστοιχούν και ε, στα όσα γίνονται στην αντιστοιχική πολιτική. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, περίπλοκο Είπε ο κ. Μασελεσί ότι υπάρχει κατακαιρματισμό ε, ε, στην κυβέρνηση του, του Καμερούν, αλλά αυτό κάνουμε και εμεί τελικά. Έχουμε διαφορετικέ πολιτικέ και δεν ε, συγκεράζονται όλε αυτέ οι διαφορετικέ πολιτικέ πάντα. Αφήστε τώρα κατά μέρο τη δική μα διαχείριση δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Χάιντι, παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω για τη μελέτη αυτή που δείχνει ότι πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία στα θέματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας και ιδίω ε, στον τομέα της ε, δασοκομείας και για τους λόγους που μας εξέθεσαν οι δύο μιλητές. Έχοντας υπόψη και το πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τα δάση, 17% πολύ περισσότερο από ό,τι συνολικά το των μεταφορών. Οδικές, ιδεδρομικές, ε, θαλάσσιες. Θα πρέπει λοιπόν να... Μάλλον οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες. Θα πρέπει να τα λάβουμε λοιπόν αυτά υπόψη, γιατί το δάσο δεν είναι μόνο ένα φυσικό αγαθό, είναι πηγή ζωή ε, και βιωσιμότητα, όπω ακούσαμε. Άρα νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να τη δράσει, δηλαδή να συντάξουμε μια έκθεση της πρωτοβουλίας, κάτι σχετικό. Αν μου επιτρέπετε κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις για συγκεκριμένα θέματα, θα δατε ίσως ότι διέρευσαν κάποια έγγραφα σε σχέση με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ιαπωνίας ε, από την Greenpeace πριν από λίγες μέρες. Και συγκεκριμένα λέγεται ότι στις δρομονές αυτές ε, το ΦΛΕΚΤ, αυτή η συμφωνία, είναι ένα σκόπελος, γιατί δεν θέλουν να ε, υιοθετηθεί οι Ιάπωνες ένας μηχανισμός που θα αντιστοιχούσε στο ευρωπαϊκό ε, φλέκτ. Και βέβαια αυτό είναι ένα πρόβλημα αν υπάρχει ελεύθερη ζώνη συναλλαγών. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και την Κίνα, τη Μαλαισία, Μαλαισία το Βιετνάμα και για τους Ιάπωνες που ε, είναι και από τις σημαντικές ε, χώρες για τις αγωγές ξυλίας. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης, πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες διαφάσεις μεταξύ ε, των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, μεταξύ των χωρών δηλαδή, που είναι αντικείμενο της μελέτης. Κύριε Βόρμς, σας ερωτώ, Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς αυτούς λογοδοσία, με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και με την καλύτερη συνέργεια του κανονισμού για την ξυλία, του FLECT και του RED+. Μήπως θα πρέπει να θετηθεί μια γενική προσέγγιση για την βάθμιση της ε, συνεργασίας με αυτές τις χώρες για να βελτιωθεί συνολικά η λογοδοσία και η χρηστή διακυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική μελέτη, όπως προείπα, και μπορούμε και εμείς να ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτά τα θέματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα στον κύριο Βάρμς για να απαντήσει και ο κύριος ε, μας έρθει στο τέλος. Σύντομα θα τα πω γιατί τα τεχνικά τα, ε, θα τα πει ο Δ. Μινάγκα. Το βασικό είναι Γνωρίζουμε ότι δεν είναι στεγανοποιημένη παρέμβαση και ξέρουμε ότι ε, θα περάσει μέσω των μικρών επιχειρήσεων. Είδαμε τι έγινε στην Νοτιοανατολική Ασία, Φιλιππίνες, φτωχότερες χώρες σε σχέση με τα Ιβάν, ε, Νότια Κορέα και Ιαπωνία. Πρέπει να βοηθά, βοηθηθούν οι Αφρικανοί εταίροι. κυρία Χάταλ ρώτησε πώς δεν θα ρίνουμε βέλτισες πρακτικές και πώς θα τις ε, περάσουμε στις άλλες χώρες. Ο κύριος Μινάκου που είναι από Δυτική μπορεί να μας πει περισσότερα. Ναι, ευχαριστώ. Κατά κάποιο τρόπο οι, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών δείχνουν ότι κάτι έχει κάνει το φλεκτ. Αυτό είναι η θετική πλευρά. Διαλέξαμε τις χώρες γιατί είχαμε στο μυαλό μας την ιδέα να δούμε αν η Γκάνα στο πέστη της δικασίας είναι απομονωμένη και σε τελείως διαφορετική φάση από την Τανζανία που ξεκινάει τώρα τη διαδικασία. Και πράγματι βλέπουμε διαφορετικά πράγματα από τη μια χώρα στην άλλη. Αν δούμε δηλαδή τη μηχανική, αν θέλετε, το φλεκτ έχει βοηθήσει τα πράγματα. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι να ενισχύσουμε τις διαδικασίες αυτές ακόμη περισσότερο. Όπως ο κ. Μαρσελεζή, στι περισσότερες περιπτώσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι Αυτό πρέπει να το κάνουμε συνολικά. Είχαμε το Καμερούν, ε, παραδείγματο χάρη, στο οποίο θετήσαμε μάλλον για το οποίο ε, εγκρίναμε κάποια μέσα. Τα εφαρμόσαμε όχι, άρα πρέπει να το δούμε συνολικά το πράγμα. Να δούμε την οπτική γωνία του φλέκτ, τι πρακτικά εργαλεία έχουμε, πώς μπορούμε να εστιάσουμε στην διαφάνεια, στην λογοδοσία. Όμως υπάρχουν και άλλες πλευρές του νομίσματος, ε, πολιτικές. Το φλέκτ τις καλύπτει αυτές τις πτυχές. Άρα Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και προσεγγίσεων. Γιατί το φλέκτε είναι άκρο πρακτικό ό,τι αφορά δηλαδή την ε, ξυλία, το πώς ε, την αξιοποιούμε, τα εργαλεία. Αλλά από την πλευρά τη πολιτική υπάρχει κενό ακόμη και κάποιε χώρες επενδύουν στον τομέα της πολιτική. Όχι και πολλέ όμω. Άρα πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό το κομμάτι της πολιτικής ευρύτερα Δηλαδή να δούμε συνολικά τη διακυβέρνηση και το ΦΛΕΚΤΑ να ασχολείται με τις λεπτομέρειες αν θέλετε σε σχέση με τη διαφάνεια. Αυτό θα ήταν μια χρήσιμη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Δεν ήξερα ότι είναι και από την Κομισιόν κάποιος εδώ και Φασουά Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Από πού είστε, από την ΤΕΦΚΟ. Μάλιστα, ορίστε. Παρακαλώ. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε και κάποια από τα δικά μου ερωτήματα. Αλλά να είμαστε και σύντομοι, δεν μα ε, έμεινε πολύ χρόνο. Τώρα μόλις πληροφορήθηκα ότι είστε εδώ. Θέλουμε την Κομισιόν να μας δώσει τη τεχνική της ε, σοφία και υπηρεγνωμοσύνη. Ευχαριστώ. Πολλά είναι τα θέματα που εθίγησαν και νομίζω ότι η διάρθρωση μεταξύ της PV και του EUTR ήταν ε, σαφής ως προς την ζήτηση και την προσφορά αυτού του προγράμματος δράσης FLECT. Θα ήθελα πάντως να επανέλθω σε μερικά σημεία της παρουσίασης για προς διευκρίνηση. Ήταν πολύ ακριβής και πολύ πλούσια η παρουσίαση Αλλά για κάποιες εταιρικέ σχέσεις με, την, με το Καμερούν, την Γκάνα ή άλλες που δεν είναι του ίδιου χαρακτήρα όπως ε, με την Αγκή του ελεφαντοστού είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το FLECT δεν είναι εργαλείο συνεργασίας ούτε χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι πρόγραμμα δράσης. Και είναι ένα πρόγραμμα δράσης που έχει δύο πτυχές, δύο σκέλη, ζήτηση και προσφορά. Υπ' αυτήν την έννοια θα συμφωνήσω πολύτως με τις ερμηνείες που δόθηκαν εδώ για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Ω προ το πρόγραμμα δράση αυτό είναι σημαντικέ λοιπόν οι συστάσει, ωστόσο να μην λησμονούμε ότι πρώτο στόχο αυτού του προγράμματο είναι να καταπολεμήσει τα προϊόντα παράνομη υλοτομία που κυκλοφορούν στην Ένωση. Αυτό εξηγεί πολλά. Ιδίω την ε, σημασία που δίνεται αυτή τη στιγμή στις εξαγωγικές εταιρείε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ως προς την ανάπτυξη και την ε, συνεργασία δεν έχουμε συνέστηση ότι η μικρή παραγωγή και οι μεσαίες εταιρείε δεν χρειάζονται και αυτές τη δική τους ιδιαίτερη προσοχή. Το δεύτερο θέμα είναι ότι στη διαδικασία μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια αξιολόγηση για τα μέσα του 2000, από τα μέσα του 2015 για να δούμε τα βασικά συμπεράσματα στα οποία διηγηθήκαμε το 2016. Πρώτον, επιβεβαιώνεται η ευστοχία του εργαλείου αυτού, του FLECT, ως προς τη διάρθρωσή του. Δεν αμφισβητήθηκε η διάρθρωσή του. Και επιτά επιμένουμε σε μια καλύτερη υλοποίηση βάσει των σημερινών ε, εξελίξεων. Βλέπουμε ότι πολλές παρατηρήσεις και συστάσεις ακούστηκαν και εδώ σήμερα στη συζήτηση. Ανάγκη παρακολούθησης και ελέγχου λόγου χάρη. Αυτό το εντοπίσαμε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας απασχολεί πολύ. Απλώς είναι τόσοι πολλοί αυτοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δράσης. Είναι τόσο δύσκολο όλοι να λειτουργήσουν στο ίδιο σχήματος κύματος. Ως προς τη συνεργασία του ΦΛΕΚ με το ΡΕΤ, εδώ έχουμε το πρόγραμμα FOE RED και σημαντικό είναι να συμβαδίσουν αυτές οι δύο διαδικασίες, αυτά τα δύο συστήματα. Προσέχουμε ιδιαίτερος όμως και τις νέες προσεγγίσεις, τα νέα εργαλεία που αναδύονται, όπως τον ΚΑΦΗ. Δηλαδή η Ευρωαφρικανική Πρωτοβουλία για την δασοκομεία λόγου χάρη που έχει ως στόχο την Κεντρική Αφρική στα πλαίσια του ΡΕΤ ή το νέο Ταμείο για την Αφρική που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Τώρα αναφέρθηκε πολύ και η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αρχίσει να σκέφτονται να οργανώσουν συνομιλίε με την Κίνα εδώ και κάποιο καιρό. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Από το 2007 υπάρχει ένα ειδικό εργαλείο που ονομάζεται BCM. Ένας ε, διμερής μηχανισμός ο οποίο ακριβώ αφορά το φλεκτ και τη συζήτηση με την Κίνα ως ε, συμμετέχουσα χώρα. Βεβαίως ε, δεν μπορώ να μην ε, παρατηρήσω ότι οι διαπραγματεύσεις κάθε είδους με την Κίνα είναι κάπως χρονοβόρες και σε καμία περίπτωση απλές. Όμως είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια συνεννόησης με την Κίνα και οδηγούμαστε όλο ένα και περισσότερο προς την κατάρτιση ενός τριμερούς διαλόγου μεταξύ Αφρικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας σε αυτό θέλουμε να καταλήξουμε, ειδικά για την Αφρική. Όμως, προς ενημέρωση, να πω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση και στάση είχε καταπιστεί και στα πλαίσια της Κόμιφακ και σε ό,τι αφορά τα δάση της λεκάνης του Κονγκό προσπαθήσαμε να πετύχουμε μια πιο ε, χειροπιαστή συμφωνία με την Κίνα για αυτές τις περιοχές της Κεντρικής Αφρικής, αλλά ε, δεν καταφέραμε τίποτα. Η Κίνα ε, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική στο να περάσει σε συμφωνίες που μπορούν να τη δεσμεύσουν οι κανόνε του παιχνιδιού αλλάζουν κάπως, διότι υπάρχει και το θέμα της καλής φήμης τη Κίνα, του καλού ονόματος που αρχίζει να έχει διεθνώ. Δηλαδή τώρα οι Κινέζοι αρχίζουν κάπως να αλλάζουν, αρχίζουν να είναι κάποιο θετικοί ω προς το να αλλάξουν τη στάση τους τα προϊόντα της Κίνας αρχίζουν να κάνουν κάπως ε, τη διαφορά με νέα πρότυπα που αρχίζουν σιγά σιγά να ισχύουν αλλά σας διαβεβαιώ ότι το θέμα αυτό βρίσκεται στην καρδιά των ε, ανησυχιών μας και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τι συμβαίνει εδώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μασελεζή να μας ενημερώσετε. Ε, είδα τότε θα μας είπατε για την Κίνα είναι πολύ χρήσιμα. Εάν θέλετε να συνοψίσετε, ναι, με συγχωρείτε, πολύ σύντομα γιατί έχω να πάω δίπλα και σε άλλη επιτροπή. Δύο σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Το μικρόφωνο σας αν θέλετε. Έσβησε. Ωραία. Ε, δύο σημεία που αναφέρθηκαν λοιπόν για την Κίνα. Πρώτον, αυτό που είδαμε στο Καμερούν. Γιατί με την αντιπροσωπή εξετάσαμε τα του Καμερούν, όχι όλη τη λεκάνη του Κονγκό. Όντω, οι σχέσει με και όντω έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κίνα είναι σε άλλο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία επαφή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα στο Καμερούν. Καμία σχέση. Και πραγματικά μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι μπορούσαμε να έχουμε ραντεβού με κάποιον από την πρεσβεία της Κίνας, όχι τον ίδιο τον πρεσβεία βέβαια, έναν εκπρόσωπό του. Ε, αυτές είναι οι σχέσεις με την Κίνα. Για το Βιετνάμ και τη Μαλαισία. στο Καμερούν παρούσα ήταν κυρίως η Κίνα διότι ακόμη και το μέγαρο των συνεδριάσεων, το παλέντε σπορ τη ε, περιοχή, οι Κινέζοι το έχουν σχεδιάσει και το έχουν χτίσει. Έτσι, ε, υπάρχει κινέζικη παρέμβαση στην αγορά με, την, ε, με τον άσχο τη παραγωγή τη Αφρική και προϊόντα που τελικά καταλήγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προϊόντα τα οποία είναι αντικείμενο επεξεργασία αυτή τη χώρα. Κίνα, Βιετνάμ και Μαλαισία. Τώρα για την παραγωγή μικρής κλίμακας, ω προ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει επιτάπητο στο θέμα. Όταν τα συζητάμε, μα λένε ότι έτσι κι αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξη που ακολουθήσαμε εμεί πρώτα στην Ευρώπη και ότι εμεί προωθήσαμε πρώτα τι μονοκαλλιέργειε με τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Οι ευρωπαϊκέ εταιρείε το θέλουν. Υπάρχει και ένα θέμα συνέπεια τη ευρωπαϊκή πολιτική εδώ. Και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Να δούμε ποια είναι τα όρια τη κοινωνική ευθύνη ε, των συνεταιρισμών που είδαμε στο Καμερούν. Και η Επιτροπή Ανάπτυξη να ασχοληθεί και με ένα θέμα που το συζητάμε επανειλημμένο, τη σχέση του business με τα human rights, των επιχειρήσεων δηλαδή και τι κάνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει όσοι πηγαίνουν να κάνουν business εκεί να σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τρίτον, νομίζω ότι η διάθεση μεταξύ του FLECT και του RBE είναι σημαντικό. Η Κίνα, η Μαλαισία και το Βιετνάμ ασχολούνται με την επεξεργασία των προϊόντων λιτομία εκτό Αφρική και μετά το Timber Beyond Forest. Δηλαδή να βλέπουμε την ξυλία και πέραν των δασών. Είναι σημαντικά σημεία αυτά. Εδώ πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει το φλεκτ προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε τους ομιλητές μας που ήρθαν εδώ και μας παρουσίασαν τη μελέτη. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μασελεσί για τα όσα μας είπε πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα θέματα από όλες τις πλευρές. Γιατί κάποιοι μου λένε εμένα ότι ο κανονισμό για την ξυλία δεν εφαρμόζεται σωστά, γι' αυτό εξετάζουμε άλλα στοιχεία, πρέπει να δούμε γιατί δεν λειτουργούν καλά και να επικεντρωθούμε και στα όσα συμβαίνουν επιτόπου, όχι μόνο στη δική μας αγορά. Θα σας ευχαριστώ και τους δύο ιδιαίτερους. Ευχαριστώ. Okay, so while we're change, while we're, um, um, I guess leaving, we can move on to item 8. Ωραία, τώρα περάσουμε στο σημείο 8, με τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της ε, ε, στην Επιτροπή του ΟΣΑΤΑΚ ε, αυτό ανέκυψε και στην προηγούμενη συνεδρίασή μα, ότι αφορά ODA, ε, ε εξωτερική δηλαδή αναπτυξική βοήθεια των επιμέρου κρατών μερών. Εξετάσαμε τι ακριβώ συνιστά ε, βοήθεια, αναπτυξική βοήθεια. Και αυτό έκανε ορισμένου συναδέλφου να ρωτήσουν πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται, ποιο πηγαίνει σε αυτέ τι συνεδριάσει, τι είδου διαβούλευση υπάρχει ποια είναι, πώς διασφαλίζεται μάλλον η διαφάνεια και λογοδοσία από πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην Επιτροπή ως ΑΝΤΑΚ. Και γι' αυτό ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει δύο πράγματα για αυτό το ζήτημα. Γιατί ακούμε συνεχώ πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση των ε, κανόνων για την άμυνα, αλλά και για άλλους τομείς, μετανάστευση, να δούμε τι ε, θεωρείται ODA και τι όχι. Έχουμε λοιπόν εδώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ για τα, κάποιες τεχνικές ε, λεπτομέρειες, για τις συνεδριάσεις, ε, τις διαδικασίες και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λίντα. Θα προσπαθήσω εν συντομία να σας εξηγήσω αφενός το ιστορικό της ε, συμμετοχής μας ε, στη ΤΑΚ και το νομικό καθεστώς που έχουμε εκεί. Αλλά θα σταθώ και σε ορισμένα ζητήματα που έχουν τεθεί επιτάπητος και επί της ουσίας ε, στην ΤΑΚ για τον υπολογισμό της εξωτερικής αναπτυξιακής βοήθειας στον ε, ιδιωτικό τομέα, στο δίκαιο παραχωρήσεων, στην ασφάλεια και το καθεξής και σε ζητήματα που ανέκυψαν σε αυτήν την Επιτροπή πρόσφατα σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση. Πρώτα δύο ιστορικά στοιχεία. Το 1960 δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή, μόλις με νέα ε, μέλη τότε, πέντε κρατημέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ηνωμένε Πολιτείε, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά. Τότε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν ένα, ένας μικρός όμιλος, ένα μικρό γκρουπ ε, χορηγών. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πλήρη ε, μέλη της ε, ΝΤΑΚ, όπως ξέρετε. Είμαστε πλήρης συμμετέχοντες, όπως ονομάζεται αυτό στον ΩΣΑ και έτσι έχουμε δικαίωμα ψήφου. Ενώ στην Επιτροπή DAC, που είναι ένα ιδιαίτερο και ανεξάρτητο μάλλον ε, τμήμα ε, του ΩΣΑ, είναι διαφορετική διαδικασία. Βεβαίω και είμαστε μέλη και εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και 20 από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Ως Επιτροπή, λοιπόν, ε, προσχωρήσαμε ως ε, χορηγός. Πολλά έχουν αλλάξει, βέβαια, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Αγώνας. Οι 20 χώρες που είναι και κάτι μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν να υπάρχει συντονισμός, γιατί για τις χώρες αυτές εμείς η Κομισιόν είμαστε εκεί ως Κομισιόν. Ε, δεν εκπροσωπούμε δηλαδή το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την Επιτροπή ε, ως χορηγό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα συντονισμού, ιδίω στο Παρίσι. Είχαμε κάποιες συνεδριάσεις για να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση, μια κοινή γραμμή όταν ε, τα πράγματα, πιο συγκεκριμένα πριν μερικά χρόνια σε ό,τι αφορά την αποδοχή συγκεκριμένων ε, ε συμβάσεων, δανειακών συμβάσεων παραχωρήσεων και αν θεωρούνταν ODA. Ε, Άλλα ζητήματα που υπάρχει κλασικά διχογνωμία μεταξύ κρατών μελών, όμω, όπω προείπα, δεν υπάρχει συνολική εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένα, ε, εμεί μάλλον, εκεί παίρνουμε το λόγο από πλευρά και εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά για την ιστορία. Εντάξει, είναι λίγο σαφή, το ξέρω. Προτιμούμε να συνεχίσουμε με αυτό το καθεστώ, γιατί αν το επανεξετάσουμε, αυτό σκεφτόμασταν, ότι η επανεξέτασή του θα ήταν μεγάλος, ε, μεγάλο ρίσκο. Γιατί μετά τη συνθήκη της Σαββόνα ε, υπήρχαν κάποιες σκέψεις για να δούμε αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πλήρες μέλος του ΟΣΑ και η απάντηση ήταν αρνητική. Επομένω, δεν θέλαμε να κάνουμε την ίδια συζήτηση στην ΤΑΚ και έτσι με ρεαλιστικό πνεύμα συνεχίσαμε ε, στην ίδια οδό. Τώρα, επί της ουσίας. Οι περισσότερες από τις συζητήσεις στην Επιτροπή ΔΑΚ και στα διάφορα επικουρικά σώματα, όπως ε, η Ομάδα Εργασίας για τα Στατιστικά Στοιχεία, είναι για το τι μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακή βοήθεια και τι όχι. Υπάρχουν ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, που υιοθετούνται συνανετικά στην ΤΑΚ και μας λένε ποιες μορφές βοήθειας μπορούν να θεωρηθούν και βοήθεια ή όχι. Τα τελευταία πέντε χρόνια λοιπόν, οι πιο σημαντικές συζητήσεις είναι μάλλον τεχνικές, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, διδανικές ε, ε, ε, συμβάσεις, μια τριετής και δύσκολη, <laughs> λίγο ε, βυζαντινού τύπου συζήτηση. Τώρα βλέπουμε ποιο είδος ε, χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξική βοήθεια και αυτές οι συζητήσεις γίνονται εκεί σε κυρίως τεχνικό και στατιστικό επίπεδο. Τώρα κάποιες φορές έχουμε και κάποια ζητήματα που είναι πιο πολιτικά. Τι μπορεί να γίνει δεκτό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και σχετική αναπτυξική βοήθεια. Και έτσι άλλαξαν, μάλλον δεν άλλαξαν πραγματικά και επίσημα, υπήρξε μια διευκρίνηση των διευθυντήριων γραμμών. Υπάρχουν λοιπόν κατευθυντήρε γραμμέ, ε, ούτε έχουν τροποποιηθεί, ούτε θα τροποποιηθούν, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση. Εμεί αυτό που ζητήσαμε, και νομίζω ότι από εκεί προέκυψαν κάποια ερωτήματα στην Επιτροπή σα, εμεί ζητήσαμε λοιπόν από την ΤΑΚ να έχουμε έναν ειδικό κώδικα για να αυξηθεί η διαφάνεια ε, των όσων δηλώνουν τα μέλη της ΔΑΚ συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επίσημη μεταξική βοήθεια. Οπότε δεν υπήρχε θέμα τροποποίηση των τεχνικών γραμμών. Απλώς θέλαμε σε έναν βαθμό να υπάρχει μια συνοχή στον τρόπο δήλωση της ε, αναπτυξιακής βοήθειας για μεταναστευτικού σκοπού. Ούτω ώστε να μην δηλώνει ένα κράτο κάτι και ένα άλλο κράτο μέλο κάτι εντελώ διαφορετικό. Ήταν για λόγου διαφάνειας λοιπόν και όπω και να έχει δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους, ε, για να αυτή τη στιγμή. Μετά. Υπήρχε ένα ζήτημα για τον τρόπο ενημέρωση των κρατών μελών για την προσέγγιση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Παρίσι. Εδώ θα θέλαμε να κάνω μια διάκριση μεταξύ των ε, τακτικών μηνιαίων ε, συνεδριάσεων της ΔΑΚ. Όλοι οι εκπρόσωποι συναντιούνται λοιπόν ε, κάθε μήνα στο Παρίσι. Τώρα αυτό δεν είναι καμία τρομερή συζήτηση, ρηξικέλευτη. Έχουμε μετά τον Ιούνιο-Ιούλιο υψηλού επίπεδου και υπουργικού επίπεδου συνεδριάσεις, ε, η πρώτη τον ιουνιο η δεύτερη τον Νοέμβριο. Και σε αυτήν την Επιτροπή και στην Κοντέρ, λοιπόν, ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο. Τι συνέβη σε υπουργικό επίπεδο και κατά πόσο θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντική αυτή η συζήτηση από πολιτικής άποψης για να ενημερώσουμε και εσά. Και βεβαίω με τα χαρά ε, σα ενημερώνουμε. Αν θεωρείτε όμω ότι πρέπει αυτέ οι ενημερώσει να γίνονται πιο συστηματικά, με τα χαρά να ερχόμαστε πιο συχνά. Ωραία, ευχαριστούμε. για τα όσα μας είπατε για τροπολειτουργία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό τον τομέα. Η κυρία Χόρμπουργκ πρώτα, παρακαλώ. those two for now, yeah. Herzlichen Dank. Maybe I... Σας ευχαριστώ. Να βάλετε ακουστικά γιατί θα μιλήσω γερμανικά. Um, Herzlichen Dank uh, für Πώς προετοιμάζετε όμως τις θέσεις και τις απόψεις σας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ποιον ε, συζητάτε προηγουμένως, ε, πώς αποφασίζετε ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των δικών σας τοποθετήσεων. Είναι οι προτεραιότητές σας, η επικαιρότητα, οι θεματικές προτεραιότητες που απασχολούν γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς ορίζετε το ότι θα συζητήσετε στην Επιτροπή Αναπτυξής Βοήθειας στην ΤΑΚ, ποια είναι τα κριτήρια. Γιατί εξακολουθώ να μην το έχω ακόμη καταλάβει επαρκώς. Επίσης μιλήσατε για το ότι υπάρχουν ε, κάποια πρόβληπτοι παράγοντες που επηρεάζουν ε, την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Εμάς ε, μας ενδιαφέρει όμως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα πολύ καλά είναι πώς ε, θα προχωρήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει στο μέλλον να συμμετέχει στην ε, χάραξη θέσης ε, την οποία θα υποστήριξετε στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας. Άρα, εσείς είπατε ότι μιλάτε μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει από εδώ και πέρα, θα στέλνουμε κι εμείς παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μήπως. Μήπως αυτό είναι μια δυνατότητα, γιατί είπατε ότι ναι ενημερώνετε για τα σημαντικά ζητήματα, αλλά εσείς αβελαμβάνετε τις αποφάσεις, ε, τι είναι δηλαδή σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε εμείς να ε, συμμετάσχουμε στην διαδικασία, λοιπόν. Γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεσμοθετήσει περισσότερο αυτή τη διαδικασία, αυτό πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Ε, στην ανταλλαγή απόψεων, για παράδειγμα, πριν το senior level meeting ή high level meeting, αν θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας, ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε τις απόψεις μας για το πώς προχωρούν οι διαδικασίες και έπειτα βέβαια να τηρούμε θα ενήμεροι για τις ε, σε εξελίξη διαδικασίες. Γιατί σας είπα ότι ε, δεν είμαστε ενήμεροι, έχουμε δύο συναντήσεις, νομίζω το senior level, το high level μία φορά μόνο, κάθε δύο χρόνια, αν δεν απατώμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και μια προφορική ερώτηση από πλευράς Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και τη δυνατότητα κατάθεσης ψηφισμάτων, αλλά εγώ νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν, να υπάρχει δηλαδή σε τακτά διαστήματα ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και σε ό,τι αφορά τις θέσεις, την τοποθέτηση να συμφωνούμε εκ των προτέρων ή ενδεχομένως να μπορεί ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει στην αντιπροσωπεία, τη διαπραγματευτική. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας της ΔΑΚ και όλης αυτής της ε, μεταρρύθμισης, νομίζω ότι θα πρέπει στην διαδικασία αυτή της διαβούλευσης να συμμετέχει περισσότερο και η κοινωνία των πολιτών γιατί και για τους κυβερνητικούς οργανισμούς ε, θα πρέπει να έχετε σε τακτά διαστήματα διαβούλευση με αυτές τις ε, οργανώσεις και θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Θα ήταν για μας πρασίνους ε, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια επιθυμία μας μεγαλύτερη διαφάνεια όπως τη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας της ΔΑΚ. Και όλα τα έγγραφα της ΔΑΚ θα πρέπει να είναι δημοσίως προσβάσιμα. Εκτός αν υπάρχει βέβαια ε, υποχρέωση εχεμήθειας. Ε, νομίζω όμως ότι για να είμαστε διαφανείς έχουμε ακόμα δρόμο. Ευχαριστώ. Η Χέιντι Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας εξήγησε την άποψή της. Αυτό που προσέξα το ενδιαφέρον, αυτό που είπατε ότι Τώρα είστε σε δημιουργές επαφές ε, για τα εργαλεία του ειδικού τομέα με κάποιες ε, χώρες. Αυτό είναι γνωστό. Ε, και είπατε βέβαια ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις σε σχέση με τη χρήση των εργαλείων του ειδικού τομέα, τη λογοδοσία και πώς μπορεί να μετρηθεί ο αντίκτυπος για να μην επανέλθουμε στις προηγούμενες καταστάσεις Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο παραπάνω για τις συζητήσεις αυτές, τι λένε οι διάφορες πλευρές, ποια είναι τα επίμαχα ζητήματα και ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα δεύτερο ερώτημα. High level panel ε, για το νόσα. Έκανε κάποιες συστάσεις για αλλαγή της εντολής πρόσφατα και για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η DAC και ζήτησε να περιλάβει και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους σε ΙΝΤΑΚ περισσότερο, να ανοίξει αν θέλετε τη συμμετοχή. Τη στηρίζει τις προτάσεις αυτές του High Level Panel Κομισιόν. Ευχαριστώ, δεν βλέπω άλλους κανείς να ζητά το λόγο, οπότε... Α, με συγχωρείτε. Κύριε βάριναν. Δεν σα βλέπω γιατί είστε εδώ στο Προεδρείο. Ναι, ευχαριστώ. Η Μαρία ρώτησε για την ε, ε επίδραση τη δουλειά του Κοινοβουλίου στη δουλειά σας ε, με του υπουργού ανάπτυξη. Τι συζητήσει έχετε δηλαδή, το Συμβούλιο πώς ε, επηρεάζει τη δουλειά σα. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Τα κράτη-μέλη δέχονται το συντονισμό πλευρά σα ή είσαστε απλώ ένα δωρητή για αυτού που κάθεται δίπλα του. Ίσως να ακούσουμε τις απαντήσεις ωστόσο για να ε, μπορέσουν και οι συνάδελφοι να ενημερωθούν καλύτερα για το μέλλον. Να συνδυάσουμε τον κατάλογο προτεραιοτήτων για να ξέρουμε τι θα ανακύψει και στο μέλλον και σε επίπεδο επιτροπή, να ξέρουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα στη διάθεσή του για να έρθει να του μιλήσει. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να απαντήσω αντίστροφα. Οι διαβουλεύσει με τα κράτη-μέλη. Όπως είπα δεν έχουμε και τόσες πολλές, διότι τα κράτη-μέλη δεν θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΤΑΚ ε, προσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Όμως, πριν από συναντήσεις υψηλού επίπεδου, ναι, έχουμε μια ενημερωτική στην Κόντεβ, είναι σε τεχνικό δηλαδή επίπεδο, δεν είναι συμβουλευτική η συζήτηση που κάνουμε. Γιατί οι περισσότερε από τι κουβέντε μα στην ΤΑΚ είναι τεχνικού χαρακτήρα. Για την ε, αναθεώρηση, τη μεταρρύθμιση στην ΤΑΚ έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ε, αναθεώρηση της δουλειάς μας από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφωνούσαμε με τις συστάσεις του πάνελ υψηλού επίπεδου και πρέπει να πούμε ότι στην ε, συζήτηση της παρακολούθησης του όλου θέματος Υπήρχαν πολύ ουσιαστικέ ε, ε, προτάσεις για μεταρρύθμιση από την γραμματεία της ΔΑΚ και οι λίγες που ήταν ριζοσπαστικές δεν έτυχαν μεγάλη στήριξη από τα μέλη. Λόγω χάρη η ψηφοφορία. Η ψήφο δεν βασίζεται πάντοτε στην ε, σύγκληση και τη συνένεση. Εδώ τα μέλη τη ΔΑΚ δεν συμφωνούσαν απολύτω. Ή το να ε, ονομάζονται και να επωνυδίζονται οι δωρητέ που δεν τα πάνε καλά ή αυτοί που τα πάνε καλύτερα από άλλου. Αυτό είναι κάτι που θεωρήθηκε προβληματικό από πολλά από τα κράτη-μέλη. Δεν ήταν υπέρ. Οπότε φοβούμε Νομίζω λοιπόν ότι αυτά που συζητήθηκαν χρήσιμα ήταν, αλλά δεν υπήρξε κάτι που ριζοσπαστικά θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργία τη ΔΑΚ. Και αν θέλετε και την άποψή μου, κρίμα. Όχι μόνο γιατί συμφωνώ και πιστεύω ότι η ΔΑΚ μπορεί να βελτιωθεί, αλλά γιατί πρέπει να δούμε και το μέλλον της στο πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας και της ατζέντα του 2030. Πρέπει να ξαναπροσδιορίσει τον εαυτό της η ΝΤΑΚ για να παραμένει επίκαιρη. Στο πλαίσιο των στόχων των, ε, της χιλιετίας, αυτό που κάνει η ΝΤΑΚ είναι ένα κλαμπ δωρητών. Και όταν συμμετέχουν και χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα ή άλλοι, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν νόημα και να το χάνουν το νόημά τους. Η ΝΤΑΚ κάνει και κάποιες προτάσεις για την δυνατότητα απότερο αποτελέσματος. Δεν ξέρω κατά πόσον η ΝΤΑΚ θα μπορέσει να προσελκύσει και νέους δωρητές. Το είδαμε και με την πρωτοβουλία όπου πρόσφατα αρνήθηκαν η Ινδία, η και άλλοι να συμμετάσχουν ακριβώς γιατί ήταν και η ΝΤΑΚ παρούσα. Κάτι το οποίο ήταν κρίμα στον ε, ιδιωτικό τομέα, επειδή είναι μια ε, συζήτηση σημαντική, εδώ συζητάμε πώς θα μετατρέψουμε και θα υπολογίσουμε τα ισοδύναμα αναπτυξιακής βοήθειας σε λόγου χάρη εγγύηση, όπως αυτές που έχουμε συζητήσει και εξηγήσει στα επενδυτικά μας προγράμματα. Εκεί Υπάρχει μια συζήτηση αρκετά περίπλοκη από οικονομικούς εμπειρογνώμονες και για τις ε, εξαγωγικές ε, ιδιαιτερότητες, τις εξαγωγικές μάλλον επιδοτήσεις. Και για να το πω πολύ απλά, η συζήτηση αφορά τα, τους συντελεστές που θα χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε την ODA, την αντιπτυξιακή βοήθεια και το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη, υψηλότερη αξίας, ε, ενώ κάποιοι, τα κράτη-μέλη, στην πρώτη κατηγορία έχουμε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία λόγου χάρη, που θα θέλαν υψηλότερου συντελεστέ ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια και από την άλλη έχουμε χώρες όπως η Αμερική αλλά και η Ισπανία ας πούμε που διστάζουν φοβερά. Διστάζουν πάρα πολύ να το επιτρέψουν. Κλασικό θέμα που επανέρχεται στην ΝΤΑΚ, το συζητάμε πολύ, ε, η ασφάλεια επίσης ήταν πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν υπάρχει συμφωνία έχουν γίνει πολλές συμβαστικέ προτάσεις από τους παράγοντες που διευκολύνουν τους facilitators, αλλά υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται ότι αυτές οι συζητήσεις θα επηρεάσουν τα των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Το θέμα είναι λοιπόν ποιο συντηρητή θα χρησιμοποιηθεί. Η διαφορά είναι μεταξύ του 3, το 4 και το 5%. Και το όλο ζητούμενο είναι ποιο ε, είναι το ποσοστό, το μερίδιο ε, μεταξύ βοήθεια που υπολογίζεται στα αναπτυξιακά συνολικά. Τέλο πάντων δεν υπάρχει συμφωνία και η Ισπανία, επί παραδείγματι, είναι από τη μία πλευρά ενώ όλα τα κάτι μέλη είναι συμπαραταγμένα από την άλλη. Τώρα το πιο κάτω μέλο ε, είναι σε κάθε στατόπεδο εξαρτάται από άλλου παράγοντε για το κόστος της αναπτυξιακής βοήθειας, πρέπει να πω ότι οι συζητήσεις δεν προχωρούν γρήγορα. Για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι η ΝΤΑΚ και ο ΙΕ συζητούν ποιο είναι το κατάλληλο ε, μέρος για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, διότι η τόστ είναι ε, ένα νέο στοιχείο και εργαλείο της αναπτυξιακής βοήθειας, οπότε κάποιοι λένε ότι αυτά πρέπει να συζητιούνται στη Νέα Υόρκη και όχι στο Παρίσι. Ως προς την ουσία όμως, η πρόοδος είναι πολύ αργή. Στόχος είναι να έχουμε κάποια προκατακτική συμφωνία πριν την υψηλού επίπεδου, αλλά αν θα τα καταφέρουμε, διότι πρόκειται για μια τελείω καινούργια έννοια που πρέπει να την ε, σχεδιάσουμε εκ του μηδενός. Πολύ αργή πρόοδος. Ως προς τις συστηματικές ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή και το να γίνονται ε, και εναλλακτικές απόψεις γνωστές, για μας δεν είναι πρόβλημα, μπορούμε να το κάνουμε Απλώς ερωτήθηκα πώς μπορούμε να το συζητήσουμε εσωτερικώς για να γίνουν σωστά οι διαπραγματεύσεις. Και πάλι όμως εξαρτάται από το θέμα. Δεν είναι και πολλές οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής ή οι υπηρεσίες της Επιτροπής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συζήτηση, αλλά υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον όταν συζητούμε ακόμη και το πού να συζητηθούν τα πράγματα αυτά, γιατί δεν συζητάμε ε, κατευθυντήριες γραμμές για τη μετανάστευση, απλώ τις στατιστικές κατευθυντήριες γραμμές. Το ερώτημα είναι πού να συζητηθούν αυτά, α πούμε, και ποιες να είναι οι γενικές διευθύνσει που θα συμμετάσχουν. Όταν συζητάμε την ασφάλεια, το συζητάμε με την ε, σχετική αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής βρίσκουμε όλες τις σχετικές υπηρεσίε για να υπάρχει μια συνεπής γραμμή, αλλά σε όλα αυτά τα θέματα μια-δυο γενικές διευθύνσεις είναι οι αρμόδιες, αλλά δεν είναι πολλές και πάλι τα κάτι μέλη σε κάποιες περιπτώσεις εκνευρίζονται, αγχώνονται και συμμετέχουν πολύ όπως έγινε με την ασφάλεια και συζητήσαμε πολύ μαζί τους. Στην περίπτωση όμως του ιδιωτικού τομέα, νομίζω μία ενημερωτική οργανώσαμε στην Κόντελ, και πάλι, επειδή το ζήτημα είναι πολύ τεχνικό όμως, περισσότερο στατιστικολόγοι συμμετείχαν για να καταλαβαίνουν το τι συζητιέται και είμαστε τυχεροί που αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της ομάδας Εργασία για τις στατιστικές είναι συνάδελφός μας. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι. και να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις στα διάφορα θέματα αλλά μετά τις επιτροπές, πριν τις συναντήσεις, μετά τις συναντήσεις, ανταλλαγή εγγράφων, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει και περώτηση. Ακόμη μια ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα επερώτησης. Για την εδραίωση της Ευρωπαϊκής άποψη και στάσει. Δεν μιλάτε με εξωτερικούς συνομιλητές. Την ε, θέση αυτή την διατυπώνεται σε επίπεδο γενική διεύθυνση ΔΕΒΚΟ, από ό,τι κατάλαβα. Μετά από συνεννόηση των υπηρεσιών και των διαφόρων ε, τμήματων. Αλλά δεν έχετε λόγο χαρδιαβουλεύσεις με την ε, κοινωνία των πολιτών, μια συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Δεύτερη ερώτηση, σημαντική για το Κοινοβούλιο να συμμετάσχουμε ανάντι σε αυτή τη διαδικασία. Και όχι απλώς να ενημερωνόμαστε ex post. Ευχαριστώ. Θα μπορούσατε να απαντήσετε, αλλά ίσως και σε επίπεδο συντονιστό να το δούμε αυτό. Να λέμε τι θέλουμε να γίνει και πώ θέλουμε να συζητάμε μαζί σα. Να δούμε πώ μπορούμε να συνεργαστούμε ή τουλάχιστον να μα δίνετε την ατζέντα τη συνάντησή σα όταν έρχεται για να ξέρουμε ποια είναι τα θέματα που θα προκύψουν. Ίσως όχι κάθε μήνα, έστω πριν την συνάντηση του Ιουλίου, με το πάνελ υψηλού επίπεδο τον Νοέμβριο και το senior level, το ανώτερο επίπεδο. Είναι ένας τρόπος να μας τα ενήμερους. Γιατί έτσι κι κάθε χρόνο κάνουμε μια συζήτηση για την επίσημη και βοήθεια. Συζητάμε τα της ΔΑΚ αλλά καλό είναι ότι τα γνωρίζουν και οι συντονιστέ και να κάνει προτάσει και η Επιτροπή μα. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Να, να πω απλώ ότι αυτό που λέτε δεν είναι καθόλου προβληματικό για μα. Απλώ ένα σχόλιο για την τελευταία ερώτηση. Δεν είναι μόνο η ΔΕΦΚΟ. Παντού στην Επιτροπή. Και σε συνεργασία με την ΑΕΔ. Κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και συζητάμε και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, διότι κάποιες φορές τα θέματα αυτά προκύπτουν στις συζητήσει. Δεν θα ήταν όμω σωστό να πω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις παρακολουθούν τι εργασίε της ομάδα εργασία περί στατιστικολογία στενά. Όταν υπήρξε κάτι να συζητηθεί με τι μη κυβερνητικέ, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να το συζητήσουμε μαζί του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πράντα και είναι πραγματικά μεγάλη η σημασία της ιστορίας που μας εξηγήσατε, του όλου ιστορικού, των πληροφοριών. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Uh, Ωραία συνάδελφοι, τώρα συζητάσουμε το σημείο 9 σε ό,τι αφορά τη συρρήκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε την έκθεση Τερέσα Χιμένεθ. Είναι εδώ η Τερέσα. Πολλές τροπολογίες έχουμε. Υπάρχουν όμω και 23 συμβαστικέ τροπολογίες τη ηγήτρια. Μπορεί να μας πει λοιπόν ε, ε, που είναι τα βασικά σημεία συμβασμού. Παρακαλώ, εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Θα μιλήσω ισπανικά. Καλό απόγευμα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει για να βελτιώσουν και ε, να συμπληρώσουν αυτό το κείμενο. Εν γέννη ε, Στόχος είναι να βελτιώσουμε τις πτυχές εκείνες που δεν μπορέσαμε να εμβαθύνουμε αρχικά ε, στην κατάσταση του κειμένου επειδή είχαμε, όπως γνωρίζετε, περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων. Θα ήθελα πάντως να αναφέρω εδώ και να τονίσω ότι πολύ επικοδομητική ε, γραμμή των τροπολογιών και να πω ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας ε, και έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες. Καταλήξαμε σε 23 συμβαστικές τροπολογίες που νομίζω ότι συμπεριλαμβάνουν, τόσο πάντων προσπάθησα ε, να συμπεριλάβω τις περισσότερες από τις ανησυχίες ε, και να αναφέρω τα προβλήματα τα οποία ε, έχετε αναφέρει, να κάνω αναφορά σε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα. Στην 13, 12 και 17 συμβιβαστική περιλαμβάνω τροπολογίες που αφορούν το ζωτικό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην κοινωνία μας και ότι στηρίζουν τη δημοκρατία. Ε, στη συμβιβαστική 4 προσπάθησα να ορίσω και να καλύψω όλες αυτές τις τροπολογίες οι οποίες εξηγούν το ευρύ φάσμα των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη συμβιβαστική 6 Μιλώ για τι αυξανόμενε απειλέ που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία των πολιτών στην προσπάθειά της ε, να επιτελέσει το έργο της. Ε, πάντοτε δεν μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζονται αυτές οι συνθήκες από την απαραίτητα ανεξαρτησία ελευθερία και ιδίω ε, βλέπουμε και κάποιες διαφορές με τον αναπτυγμένο κόσμο στην συμβιβαστική πρόταση 7. Αναφέρω συγκεκριμένα ποιες απειλές αντιμετωπίζουν οι ακτιβιστές. Στην 13 συμβιβαστική πρόταση περιλαμβάνω τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες μιλούν για τις στρατηγικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις για να περιορίσουν την επιρροή της κοινωνίας των πολιτών δηλαδή να επιβαρύνουν με γραφειοκρατικές διαδικασίες που δυσχεραίνουν το έργο τελικά των ΜΚΟ, στερώντας τους την ευελιξία και την ταχύτητα δράσης στη συμβιβαστική, για να μην ε, μπορούν δηλαδή τελικά να επιτελέσουν το έργο τους ε, ως θέλουν. Στην 18 μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, για τα συνδικάτα και για τις σχέσεις τους με την κοινωνία των πολιτών και πώς μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι φορείς για να προσπίσουν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να υπάρξει καμία κατάχρηση. σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα ή κάποιο άλλο, κάποια άλλη πλευρά. Στην 23, συμβιβαστική πρόταση, λέω ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις διμερείς ε, σχέσεις για να είναι εγκυμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να περιλαφθεί η λεγόμενη θετική αιρεσιμότητα. Λίγο πολύ αυτά πολύ συνοπτικά, τηλεγραφικά. Αύριο, μια μισή μεσημέρι, θα έχουμε την πρώτη συνάντηση με τους κοιόδης συζητητές. Ήδη έχω λάβει το input ορισμένων συναδέλφων, νομίζω όμως ότι... Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Με τα περισσότερα μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στόχο είναι να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και είμαι σχεδόν βεβαία. Γιατί από τότε που ξεκίνησα να επεξεργάζομαι αυτή την έκθεση, από όλε τι πλευρέ δεν έχω λάβει παρά υποστήριξη. Ουσιαστικά ε, όλοι είπαν ότι με το πνεύμα της έκθεσης είναι σύμφωνοι. Επομένως, και επειδή είναι και έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε την μέγιστη δυνατή υποστήριξη στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή αλλά και συνολικά στο Κοινοβούλιο ώστε να έχουμε ισχύ, να έχουμε δύναμη και η έκθεσή μας να ληφθεί υπόψη και να έχει κάποιο, κάποια χρησιμότητα, κάποιο όφελος. Όλοι νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας να δείξουμε την απαραίτητη βούληση για να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φρουντζούλικα. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε την ε, εξωσορροπημένη αυτή έκθεση και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Είναι θεμελιώδης σημασία αυτή η έκθεση για να δείξουμε την αυξημένη διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών και της κοινωνίας των πολιτών και του χώρου που κατέχει. Μέσω των τροπολογιών που κατέβαλα κατέθεσα, ήθελα να δείξω ότι δεν είναι μόνο οι αναπτυσσόμενες χώρες που ε, συρρυκνώνουν αυτόν τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς συμβαίνει ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα συνολικό και παγκόσμιο φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να διατηρήσει την αξιοπιστία τη, εάν δεν αναγνωρίσουμε και εμεί δηλαδή ότι και εμεί έχουμε αντιμέτωποι με τέτοιου είδου προκλήσει. Ήθελα επίση να επισημάνω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι και αυτά σημαντικά, ε, καθώς και οι κυβερνήσεις για τον διάλογο και την ε, συνεργασία από όλες τις πλευρές. Τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και όταν συνεργάζονται με την κοινότητα των πολιτών, με τον ιδιωτικό τομέα, με τα κόμματα τη αντιπολίτευση, τι αρχέ της ε, τοπική αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να διατηρούν έναν ανοιχτό χώρο για την κοινότητα των πολιτών. Πρέπει να ενισχύσουμε τη στήριξή μα για την πλήρη συμμετοχή των μειονοτήτων, ε, συμπεριλαμβανομένων και των ηθαγενών και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε πολιτισμικές, κοινωνικές και άλλε ε, ε, πολιτικές διαδικασίες. Μηχανισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων και των ε, ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, με τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να ενισχυθούν και να ενισχυθεί και ο ρόλο των φορέων τη κοινωνία των πολιτών. Ε, επισημαίνουν την, συμφω... την σημασία τη ε, περιφερειακή συνεργασία σε αυτόν τον κλάδο και θεωρώ ότι θα πρέπει να παροτρύνουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε να προωθούν ε, τις βέλτιστες πρακτικής, του διαλόγου και της ε, προστασίας και της ε, συμπερίληψης της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία νότου-νότου είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί κάποιες χώρες έχουν δείξει και έχουν δραματίσει ηγετικό ρόλο και έχουν αποτελέσει παράδειγμα και για τις γειτονικές τους χώρες. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των επιχειρήσεων. Ο ιδιωτικό τομέας είναι ένα βασικό εταίρος στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην ασφάλεια ανεφοδιασμού, δέουσα επιμέλεια και το καθεξής, αλλά και ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το συνδικαλιστικό κίνημα. Ε, Συγχαίρω και πάλι την εισηγήτρια και ελπίζω να καταλήξουμε στη συμφωνία για αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο. Ευχαριστώ, Μαρία Χόιμπουκ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Τερέσα για τη δουλειά της ε, και πάνω στην έκθεση αυτή και στη... για τις ε, πολλές συμβαστικές ε, τροπολογίες που έχει καταρτήσει ό,τι αφορά τη σημασία της έκθεσης. Νομίζω ότι πραγματικά είμαστε όλοι σύμφωνοι και σίγουρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ένα μεγάλο κομμάτι της των πολιτών και επιρροή της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να μιλήσουμε για δημοκρατικές κυβερνήσεις. Ε, συνολικά οι πράσινοι ε, συμφωνούμε με τις περισσότερες ε, τροπολογίες συμβιβαστικές. Ε, δύο σημεία θέλω να επιμείνω όπου θεωρώ ότι οι προτάσεις της εισηγήτριας δεν μας εκπροσωπούν επαρκώς. Το πρώτο είναι σε ό,τι αφορά την ευθύνη του ιδιωτικού τομέα και το δεύτερο θέμα είναι τι γίνεται εντός Ευρώπης. Ε, πρώτον, σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά ο ιδιωτικό τομέας είναι σημαντικός ε, και έχει ε, πολλά να συνεισφέρει και στους, στις βιώσιμες και στους αναπτυξιακούς στόχους. Δεν τίθεται αυτό υπό αμφισβήτηση. Το θέμα είναι δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα πολλές φορές μπορεί ε, να είναι προβληματικές και ρηψοκίνδυνες. Γι' αυτό λοιπόν σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να μπορέσουμε να εισαγάγουμε τους απαιτούμενους ε, μηχανισμούς ώστε να μπορούμε να έχουμε λογοδοσία ε, και σε ό,τι αφορά να το αφήσουμε αυτό εθελοντικό νομίζω ότι δεν είναι κάτι θετικό και σε ό,τι αφορά τα περιθώρια που και το χώρο της ε, κοινωνίας των πολιτών. Πολλές φορές ακούμε περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις, ε, στους ακτιβιστές ε, προσπαθούν να τους αποθαρρύνουν. Παραδείγματο χάρη, παρενοχλήσεις, μέχρι και άσκηση βίας. Έχουμε διαβάσει τέτοιες αναφορές, γνωρίζουμε. Μάλιστα περιπτώσεις που υπάρχουν και απειλές για απειλές κατά της ζωής ε, των ακτιβιστών. Και ό,τι λέμε εμείς πολλές φορές πέφτει στο κενό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν ε, πολύ ριζοσπαστικό εδώ να υπάρχουν κάποιοι δεσμευτικοί κανόνες, αυτό να προτείνουμε, γιατί νομίζω ότι είναι λογικό αίτημα ε, σε σχέση με όσα παρατηρεί κανείς να συμβαίνει. Γιατί αν αφήσουμε στον ιδιωτικό τομέα το, την ευθύνη τότε νομίζω ότι δίνουμε αρνητικά κίνητρα και στέλνουμε και λάθος μηνύματα. Επομένως, ε, ε, σίγουρα χρειάζεται μια ισχυρή διεθνή συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα για να ρυθμιστεί ε, αυτό το ζήτημα, για να δείξουμε ότι τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες παιχνιδιού που να ισχύουν για όλους. Και αν με επιτρέπετε σύντομα για την Ευρώπη, ε, και τα περιθώρια που έχουμε εδώ. Ε, στην Επιτροπή μας πριν από ένα μήνα νομίζω είχαμε μια συζήτηση και πολλοί συνάδελφοι από διαφορετικές πολιτικές ομάδες ε, είχαν ζητήσει και σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών να συζητήσουμε για τα περιθώρια και το χώρο που θα έχει η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι πολύ ε, λογικά μπορούμε να το αιτιολογήσουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος για να το περιλάβει αυτό. Ίσως θα πρέπει στη διάσκεψη των πρώτων ε, των επιτροπών να συζητηθεί. Γιατί είναι ένα επίκαιρο θέμα, καυτό θέμα και θέλουμε να καλυφθεί. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ακριβώς ε, η εισηγήτρια πώς επιθυμεί να ρυθμίσει αυτά τα θέματα σε σχέση με το τι γίνεται εδώ στην Ευρώπη δηλαδή. Δεν νομίζω ότι καλύπτεται θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και όχι ε, να κοιτάμε τι γίνεται στο βορρά στο νότο και τα του οίκου μας να τα αφήνουμε εκτός. Πρέπει και τα του οίκου μας να ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ. Σασάριο Μπέντο. Από τη Γενική Διευθυντή Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και χαιρετίζουμε πολύ ε, αυτή την έκθεση. Είναι ιδιαίτερα επικαιρή γιατί έχει να κάνει με ένα από τα πιο κέρια ζητήματα ε, που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι φορεί τη κοινωνία των πολιτών και αναγνωρίζει και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί ήδη για τη στήριξη τη κοινωνία των πολιτών. Εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο τη προσοχή η κοινωνία των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ε, και δυναμική ε, σε ό,τι αφορά την άλυψη δράση ε, για να αντιστρέψουμε την πορεία συρρήκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε και την έκθεση για την κοινωνία των πολιτών στι 28 Απριλίου που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναδεικνύει όλη τη δουλειά που έχει γίνει μετά την υιοθέτηση τη ανακοίνωση για την κοινωνία των πολιτών στι χώρε εταίρου του 2012. Την περασμένη εβδομάδα, ή μάλλον αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα στις 19 Ιουνίου, το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα όπου επανεπιβεβαιώνει και πάλι την ε, προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και εκφράζει σημαντικές ανησυχίες ό,τι αφορά το συρρυκνούμενο χώρο της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές χώρες και ε, τονίζει και τη σημασία για τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Η συνέντευξη που έχει επιτευχθεί ε, επιβεβαιώνει εκ νέου την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού και συμπεριληπτικού χώρου για την κοινωνία των πολιτών με ε, δημοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα στο φορά τελείωση αποφάσεων και η έκθεση αυτή είναι πολύ καλογραμμένη και δείχνει ξεκάθαρα και τη θέση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το σημαντικό αυτό θέμα. Σα ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ και ο κύριος Ρώση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα είπε η συνάδελφος από την DG DEFCO. Αναφέρθηκε σε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις, ιδίω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που επιβεβαιώνουν εκ νέου την ξεκάθαρη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ε, για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στην εξωτερική της δράση. Επομένως και εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε. Τερέζα, θες και πάλι τον λόγο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση και για τις επισημάνσεις του συμφωνώ με αυτά που είπαν οι σκιώδεις. Και όταν λέτε για την Ευρώπη, ότι δεν αναφέρουμε την Ευρώπη, δεν συμφωνώ. Στη 12 συμβιβαστική τροπολογία συγκεκριμένα λέμε worldwide. Όταν μιλάμε για την κοινότητα των πολιτών, πρέπει την κοινότητα των πολιτών να τη δούμε σφαιρικά. Και πάνω ε, με αυτό το πνεύμα έχω συντάξει τις ε, τροπολογίες. Δηλαδή δεν θέλω να εστιάσω σε συγκεκριμένες χώρες, ή ε, χώρες ευρωπαϊκές ή όχι, γιατί φυσικά και λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες χώρες. Μην χάσουμε την δυνατότητα να αναφερθούμε. Το λέμε και στη συμβιβαστική, αλλά γενικά μιλάμε. Μιλάμε για local strategies επίσης. Αλλά και πάλι υπάρχουν πολλές άλλοι, πολλές άλλες διατυπώσεις που είναι πιο γενικόλογες. Εμείς προσπαθούμε απλά να εστιάσουμε σε αυτό που είναι το αντικείμενο τη έκθεσης. Δεν είμαστε Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών, είμαστε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Εγώ εργάζομαι και στην ΛΥΠΕ και είναι και η επίσης που ασχολείται με το θέμα και συμφωνεί με τον τίτλο που λέτε εσεί να τον αλλάξουμε. Υπάρχουν πολλέ οργανώσεις που θέλουν πραγματικά σε αυτό να εστιάσουμε. Όπως το λέμε στη 13 συμβαστική η εμφυλιβία, οι αυθαίρετες κρατήσεις, λογοκρισία, ο περισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Και όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, απευθυνόμαστε στις κυβερνήσεις, αλλά και όχι μόνο στους κρατικούς φορείς, και στους μη κρατικούς φορείς αναφερόμαστε, όταν αυτοί θέλουν να περιθωριοποιήσουν ε, τη φωνή της των πολιτών. Νομίζω λοιπόν δεν ξέρω πώ θέλετε να κάνουμε μια άλλη έκθεση για συγκεκριμένε χώρε. Να το κάνουμε. Μπορούμε να συντάξουμε μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία. Αλλά νομίζω ότι καλά τα έχουμε ορίσει, έχουμε εργαστεί πολύ αρμονικά και αν βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα μπορούμε να τα ξαναδούμε. Στην αυριανή, όπως είπα, συνάντηση με τους κοιόδες εισηγητές θα το κάνουμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαι ανοιχτή σε όλες τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου την εισηγήτρια. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και είμαι βέβαια ότι θα προλάβουμε πριν τις διακοπές να έχουμε μια συνεννόηση. 30 Αυγούστου θα ψηφίσουμε. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο για σήμερα, σημείο 10, ώρα των ερωτήσεων. Ερώτηση προς εμένα την ίδια. Δεν θα διαβάσω την ερώτηση, αφορά την, τον λοιμό και την ανθρωποστική κατάσταση επίγουσα κατάσταση σε πολλές αφρικανικές χώρες και την Ιεμένη. Οι ειδήσει που ακούμε από τις χώρες αυτές για το γεγονός ότι η βοήθεια δεν φτάνει εκεί που πρέπει. Η κυρία Ανδρούλα Καμινάρου είναι εδώ μαζί μας νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ελπίζω να μας ενημερώσετε. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη Σομαλία και, το Σομάλιλα, και τη Σομάλιλαντ, αλλά... αλλά θα περιμένω να ακούσω εσάς πρώτα. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το μικροφωνό σας για τη διερμηνία. Ευχαριστώ. Θα δείξω αρκετά ζητήματα που αφορούν τις περιπτώσεις λοιμού, απλώς πολύ γρήγορα. Από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, τότε μιλήσαμε για το γεγονός ότι υπήρχε υποχρηματοδότηση από όλους τους δωρητές αυτό το διάστημα. Τι έχει γίνει λοιπόν εντωμεταξύ. Από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενέτεινε την χρηματοδότηση ως απόκριση στην ε, κατάσταση λοιμού και ένα τρίτο των αναγκών για την ώρα έχουν χρηματοδοτηθεί. Όπως είχα πει, το πρόβλημα με την απόκριση στους λοιμούς δεν είναι μόνο θέμα χρηματοδότησης, αλλά είναι θέμα και πραγματικής προσφοράς επιτόπου βοήθειας, της αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτίων του λοιμού, των γεωγραφικών προεκτάσεων. Θα σχολιάσω πώς επηρεάζεται η όλη περιοχή από αυτά και η ανάγκη περισσότερου συντονισμού και συνεργασίας όλων των φορέων επιτόπου. Θα σας ενδιέφερε να μάθετε πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ε, προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν τους λοιμούς. 668 εκατομμύρια το 2017 και μόνον ως τώρα. 300 είναι ανθρωπιστική βοήθεια και 370 ανάπτυξη. Η διαίρεση μεταξύ των τεσσάρων περιπτώσεων λιμών είναι ως εξής. Η Εμένη 116, Νότιο Σουδάν 146, Σομαλία 119 και Σομαλία 217. Πρέπει βεβαίω να δούμε και τις γεωγραφικές προεκτάσει όταν μιλάμε για λαιμού. Λόγω χάρη το Νότιο Σουδάν και η περίπτωση του λοιμού στο Νότιο Σουδάν σημαίνει 2 εκατομμύρια Νότιο-Σουδανοί να φεύγουν στις γειτονικέ χώρες. Αντιδρούμε λοιπόν και στις ε, παρελκόμενες, συνέπειες του λοιμού. 347 εκατομμύρια ανθρωπιστική ε, απόκριση λοιπόν στις ε, χώρες για τους οποίους συζητούμε και τους πρόσφυγες μαζί που φεύγουν από αυτές τις χώρες. 200 στη, στο Νότιο Σουδάν, 205 ε, στην, στο κέντρο της Αφρική και 105 στο Τσάντ. Εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε προσπαθήσει για αυτούς τους λοιμούς να έχουμε ένα συνολικό ποσό και καταλήξαμε στα 736 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη. Εάν προσθέσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τα κράτη-μέλη, η συνολική συμβολή για τους τέσσερις λοιμούς είναι 1,4 δις. 1,4 δις που είναι περίπου το 60% όλης της ανθρωπιστικής απόκρισης που θα διατεθεί στην περιοχή. Δεν είναι και λίγο. Αξισημείωτες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη. Απλώς, σύντομα, να αναφερθώ στην Ουγκάντα, όπου ήμουν εκεί την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας, διότι υπήρχε μια σύνοδος κορυφής για την αλληλεγγύη προς την ε, Ουγκάντα, με προσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Επιτρόπο Στυλιανίδη, ο οποίος εκ μέρους του αυτού του και εκ μέρους του Επιτρόπου Μίμητσα μίλησε για 5 εκατομμύρια. 85 εκατομμύρια για την ανάγκη ε, να περιθάλψει η Ουγγάντα τους νοτιοσυδανούς ε, πρόσφυγες. Πέρσι 800.000 ε, νοτιοσουδανοί διέφυγαν στην Ουγγάντα. Σε αυτήν την σύνοδο αλληλεγγύης 350 356-358 εκατομμύρια δολάρια ε, δεσμεύτηκαν για να αντιμετωπίσει η Ουγγάντα την κρίση των προσφύγων, δύο τρίτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διέρεση 95 εκατομμύρια σε δολάρια, 85 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ 95 δολάρια και 195 τα κρατη μέλη. Εάν δούμε τι υποσχέσει των υπολείπων, τι δεσμεύσει των υπολείπων δωρητών, είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Καναδά, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Κατάρ, η Ιαπωνία έχουν 10 εκατομμύρια. Μετά η Νότια Κορέα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αυστραλία και η Νορβηγία 5. Η Ινδία, αλλά και μικροποσά από τις Αφρικανικές χώρες Γκαμπών, Κένια, ε, Σομαλία η οποία και αυτή προσφέρθηκε να βοηθήσει την Ουγγάντα να καλύψει τις ανάγκες των Νότιο Σουδανών, Κίνα, μόνο μισό εκατομμύριο. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε αυτές τις ειδικέ περιστάσεις, που είναι τελευταία εξέλιξη η προστασία των Νοτιοσουδανών στην Ουγγάντα, βλέπουμε ότι και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συν τα κράτη-μέλη, δίνουν τα δύο τρίτα της συνολικής βοήθειας, απόκρισης ως προς την εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους λοιμούς και σε σχέση με το τι είχε δεσμευτεί αρχικά. Εάν πάρουμε την περιοχή του Τσάντ το Φεβρουάριο, 105 εκατομμύρια είχαμε δεσμεύσει, εκ των οποίων 90 προς την Ιγυρία, στο κέρας της Αφρικής. Αρχικά προβλέπαμε τον Φεβρουάριο 82 εκατομμύρια. Τον Μάρτιο φτάσαμε τα 165, εκ των οποίων 100 για τον Νότιο Σουδάν και 65 στην Σομαλία, την Αιθιοπία και την Κένια. Για την Ιεμένη, τον Απρίλιο η Επιτροπή ε, ανακοίνωσε επιπροσθέτως 17 εκατομμύρια. 70 εκατομμύρια. Ε, στην αρχή της χρονιάς ε, αυξήσαμε το ποσό για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Το άλλο που θέλω να αναφέρω είναι ποιος άλλος αντιδρά στους λοιμούς. Πως άλλοι διεθνείς δωρητές έχουν συμμετάσχει. Για την Ιεμένη η συνεισφορά των έξω ευρωπαϊκών δωρητών 350 εκατομμύρια, εκ των οποίων 85% από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Νότιο Σουδάν, οι εξωευρωπαϊκοί δωρητές, 760 εκατομμύρια, εκ των οποίων μεγαλύτερος δωρητής ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη Σομαλία το ίδιο, 300 εκατομμύρια από εξωευρωπαϊκούς, τα μισά από, τις, από την Αμερική, στην Ιγυρία 270, εκ των οποίων μεγαλύτερος δωρητής από όλους είναι οι Αμερικανοί. Νομίζω αυτά είχα να πω τώρα και αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι. Έχω εγώ ένα ερώτημα, πιο συγκεκριμένα για τη Σομαλία. Πιο συγκεκριμένα για το Σομάλιλαντ. Έχουμε πολλούς ομογενείς ε, του Σομάλιλαντ στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Κάποιοι επέστρεψαν από το Σομάλιλαντ πρόσφατα και ε, μου μετέφεραν εικόνες ε, του Ρωμερού Λιμού και ξεσπάσματος χολέρας. Ξέρετε ότι πρόκειται για μια ε, ανεξάρτητη οντότητα εντός του κράτους της Σομαλίας, αλλά δεν αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος, παρόλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης του. Και η βοήθεια δεν φτάνει μέχρι εκεί. Οπότε, εντάξει, δίνουμε τη βοήθεια στη Σομαλία, αλλά πώς είμαστε σίγουροι ότι φτάνει όντω εκεί που πρέπει. Ελέγχεται δηλαδή αν φτάνει η βοήθεια τελικά στο Σομάλιλαντ και το ίδιο ισχύει και για τι υπόλοιπε χώρε. Σε κάθε χώρα υπάρχει συγκεκριμένη και λεπτομεριακή ανάλυση ε, για τις ανάγκες που καλύπτονται ε, και πιο συγκεκριμένα για τη χολέρα, στη Σομαλία ευρύτερα. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι περίπου 50.000 έχουν ε, ασθενήσει κυρίως ε, στην Ήπεθρο, αλλά και ευρύτερα στην επικράτεια της Σομαλίας. Στο Σομάλιλαντ ξέρουμε ότι υπάρχουν κρούσματα χολέρας. Ήδη εξετάζουμε πώς ε, θα ανταποκριθούμε σε αυτό το φαινόμενο και έχουμε ένα πρόγραμμα 4,5 εκατομμυρίων ε, με τη UNICEF για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Παρακολουθούμε λοιπόν του συναγγεί, ε, τι ανάγκες και ανταπακρινόμεθα αναλόγως. Τώρα, για τη χολέρα και πάλι στην Αιθιοπία. Και εκεί υπάρχουν όλα ένα και περισσότερα κρούσματα χολέρας και μηνύματα που μας δείχνουν ότι ε, επιδεινώνεται η κατάσταση. Όμως, σε ό,τι αφορά την Αιθιοπία. Ε, δεν αποκαλείται ξέσπασμα χολέρας ε, το φαινόμενο, ε, αλλά ε, οξίας διάρειας. Δώσατε πολλά στοιχεία, λέει Πρόεδρος, μπορείτε ίσως να μας τα στείλετε και σε μένα και στην γραμματεία, γιατί και οι συνάδελφοι θέλουν να γνωρίζουν. Βλέπουμε ότι μόνο το 1 τρίτο των αναγκών ουσιαστικά καλύπτεται. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί μόλι το 1 τρίτο των αναγκών καλύπτεται. Και μετά, γιατί το αποκαλούν διαφορετικά δηλαδή στην Αιθιοπία, γιατί δεν το λένε χολέρα. Και για τη Σομαλία, στο Σομαλιλάντ. Σα τα λέω όλα μαζί για να απαντήσετε από κοινού. Μπορεί να μην το έχετε εύκαιρο αυτό το στοιχείο, αλλά θα ήθελα να μάθω πού πηγαίνει η χρηματοδότηση. Ε, διοχετεύεται μέσω ΜΚΙΟ, γιατί η κυβέρνηση δυσκολεύεται πολύ ε, να συνεργαστεί με τους παγκόσμιους οργανισμούς, γιατί δεν ε, είναι αναγνωρισμένο κράτος. Πώς λοιπόν διανέμεται η χρηματοδότηση για να φτάσει εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από άλλα μέλη. Όχι. Παρακαλώ, απαντήστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το πώς ε, διοχετεύονται οι πόροι. Ε, διάφορες ΜΚΟ ε, σε αυτή την περιοχή έχουν πρόσβαση στον πληθυσμό. Εμείς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν αυτή τη βοήθεια υπάρχει συμφωνία ότι μπορεί να η βοήθεια σε όλη την επικράτεια της Σομαλίας, αλλά είναι βέβαιο ότι κάποιες είναι πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Ωστόσο, και στη Σομαλία και στο Σομάλιλαντ, αν θυμάμαι καλά, νομίζω μέσω του Ερυθρού Σταυρού έχουμε πρόσβαση σε αυτό το τμήμα της χώρας. Υπάρχει όμως πολύ συγκεκριμένη χαρτογράφηση για το ποιος έχει πρόσβαση σε κάθε περιοχή και ποια ανάγκη καλύπτεται κάθε φορά, αν πρόκειται για τροφή ή κάτι άλλο. Ακολουθούμε το σύστημα OTSA για να το κάνουμε αυτό. Στη Σομαλία είναι ιδιαίτερα περιπλοκή κατάσταση και πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Έχουμε μια ομάδα περίπου 40 ΜΚΟ υπό ε, τη διαχείριση ότσα και κυβέρνησης για αυτή τη χρηματοδότηση. Για να εντοπίσουμε ακριβώς τα κενά και να συγκορευτούμε ότι θα φτάσει τελικά αυτή η βοήθεια σε αυτούς που το χρειάζονται. Μόλις το 1 τρίτο της ανταπόκρισης ε, διατίθεται τελικά. Αυτό είναι πρόβλημα εφόσον δεν έχουμε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, εφόσον σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και συνεχίζονται, συνεχίζονται συγκρούσεις. Στην Ιγερία, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε ε, το ποσό που ε, προβλέπεται σε καθένα από αυτούς τους Αν είχαμε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές και είχαμε τη δυνατότητα να τα δώσουμε παντού, θα ήταν καλύτερα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά εφόσον υπάρχουν ζητήματα και δεν έχουμε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, γιατί συνεχίζονται συγκρούσεις, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Αλλά τα στοιχεία είναι καλύτερα από αυτό, από την εικόνα που διαφαίνεται και για τις συγκρούσεις έχουμε περίπου 30-50% γιατί με τις ε, πρόσφατες υποσχέσεις ε, αυτό διακυμαίνεται. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω εδώ. Για την επιστηστική βοήθεια, για παράδειγμα, προσπαθούμε να σιγουρευτούμε ότι όπου αυτό είναι δυνατόν, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης του εισοδήματός του για να μην εξαρτάται συνεχώς από την ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ιγυρία, για παράδειγμα, ο ΦΑΟ διανέμει ε, σπόρους σε εκατομμύρια ε, ανθρώπων για να μπορούν να τους καλλιεργήσουν και ταυτόχρονα βέβαια τους ε, χορηγείται και τροφή για να μην μπουν στον πειρασμό να φάνε τους πόλους αντί να τους ε, σπείρουν. Επομένως, ταυτόχρονα, όπου αυτό είναι δυνατόν, τους στρέφουμε και τους δίνουμε και τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν, τους ώστε κάποια στιγμή ε, να ξεφύγουν από αυτή την σχέση εξάρτησης από την ανθρωπιστική βοήθεια. Κάτι άλλο που κάνουμε και όλα αυτά που ανέφερα έχουν σχέση και την αναπτυξιακή βοήθεια και τα όσα κάνει. Εμείς συνεργαζόμαστε πολύ στενά για να δούμε που σταθεροποιείται η κατάσταση, που υπάρχουν περιοχές όπου ο κόσμος μπορεί να επιστρέψει στα χωριά του και τότε θα έχουμε χρηματοδότηση ανοικοδόμησης αν θέλετε των υποδομών που ενδεχομένω έχουν πληγεί, σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Επομένω, τα εξετάζουμε και λίγο πιο μακρόπνοα το όλο θέμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μα στείλετε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, πολύ χρήσιμο και ιδίω για, για την ε, περιοχή αυτή τη Σομαλίας, τη Σομάλιλάντ, που μα ενδιαφέρει όλο ιδιαίτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε και να ζητούμε από τους υπουργού μας ε, λόγο για το τι κάνουν. Για να παρακολουθούμε την κατάσταση. 11 διάφορα, δεν έχω κάτι εγώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη συνεδρίαση 12 Ιουλίου. Όχι, με συγχωρείτε τη Δευτέρα στις 7.30 στο Στρασβούργο και μετά ψηφοφορίες και μετά 12 Ιουλίου. Ολόκληρη τη μέρα και 30 Ιουλίου, λέει πρόοδο, μόνο το πρωί. Σα ευχαριστώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο.